No, si lo sé, por eso vamos, vamos a empezar ya, porque si no... Bueno, buenos días a todos. Καλημέρα σε όλους. La sesión de hoy. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Hoy el, el, el punto 7. Que... Είχαμε αφήσει σε κρεμότητα από χθε το σημείο υπαριθμών 7 για την τροποποίηση του κανονισμού 1198 του 2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Λίας. Η έκθεση αυτή την είχε αναλάβει ε, η ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Φερέιρα, αλλά επειδή ο κύριος Φερέιρα είναι στην συνεδρίαση των χωρών ΑΚΕ, δεν μπορεί να παραστεί και να παρουσιάσει την έκθεσή του και έχει αναθέσει στην κυρία ε, Φιγκερέιντο να ε, παρα, παρουσιάσει την έκθεσή του. Να σας δώσω το λόγο. Θέλετε να λάβετε το λόγο τώρα ή να δώσετε το λόγο στην Κομισιόν μετά πρώτα. Θέλετε πρώτα να μιλήσετε εσείς ή να δώσετε το εσεί η κυρία Φιγκυρέιντο. Όντως, μέσα σε αυτή την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Όντω για αυτή την έκθεση μάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αιτιολόγησε την πρότασή της Παρουσίασε βεβαίω ένα έγγραφο με μια πρόταση, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να παρευρεθεί εδώ κάποιο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα αιτιολογήσει, να μα παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Αυτό περίμενα εξάλλου. Ε, γιατί ο εισηγητής ε, κρίνει ότι μπορεί γενικά να γίνει αποδεκτή η πρόταση εκτός από κάποιες συστάσεις με στόχο να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές αναθεωρήσεις αυτού του κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει την πρόταση του κ. Φερέιρα και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να παρουσιάζει τη θέση της. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση που έχετε ενώπιόν σας είναι μία ακόμα απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσπαθήσει να μετριάσει τις επιπτώσεις της παρούσας οικονομικής κρίσης. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη πρόταση για την τροποποίηση του Ταμείου Αλίας, αλλά εκ παραλήρου με αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε παρέμοιες προτάσεις τροποποίησης και για άλλα ε, διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία συνοχής, τα γεωργικά διαρθρωτικά ταμεία και σε όλες τις περιπτώσεις ο στόχος είναι κοινός. Όπως γνωρίζετε, η ανάγκη να μετριαστούν τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης ε, είναι άμεση για πολλά κράτη-μέλη, ιδίως για κράτη-μέλη που επιβάλλονται ε, προγράμματα λιτότητας και μας ενδιαφέρει η καλύτερη διαχείριση των πολιετών προγραμμάτων, διότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας ε, σε διοικητικό επίπεδο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ε, τα προγράμματα τα οποία υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, επαναλαμβάνω εκ παραλίλου με τα όσα προτείνουμε και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ταμεία, είναι να επιλύσει το πρόβλημα της ρευτότητας μέσω μιας τροποποίησης η οποία προτείνει περισσότερη ευελιξία ώστε να μπορεί να πληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο γρήγορα μεγαλύτερες ποσότητες χρημάτων ε, από τα κονδύλια που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ώστε να έχουμε μία ένεση κονδυλίων στις χώρες οι οποίες ε, απαιτούν κονδύλια και να είναι και μια μορφή υποστήριξης, ε, να μπορούν να κυκλοφορήσουν τα κονδύλια, να μπορούν τα κράτη-μέλη να δώσουν στους δικαιούχους ε, περισσότερα κονδύλια για την υλοποίηση των προγραμμάτων και αυτό που κάναμε ήταν να προτείνουμε ένα σύστημα στο οποίο αυξάνεται κατά 10% η συγχρηματοδότηση, το ποσοστό συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας με στόχο τα κράτη-μέλη από εκεί και πέρα να μπορούν να ζητήσουν μεγαλύτερη πληρωμή από τα κονδύλια τα οποία θα ελάμβαναν υπό αμαλά συνθήκα. Αυτό δεν αφορά όλα τα κράτη-μέλη, επαναλαμβάνω, αλλά μόνο τα κράτη-μέλη τα οποία ε, έχουν ε, κάποιο από τα προγράμματα υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για τις χώρες του ευρώ ή το ισοζύγιο πληρωμών για τις χώρες που βρίσκονται εκτός ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι την πρόταση αυτή μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν έξι κράτη-μέλη τα οποία υπάγονται σε αυτούς τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Λιτωνία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Ο στόχος είναι, όπως σας έλεγα, να αυξηθεί το ποσό που δίνεται από κοινοτικά κονδύλια και που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επισημάνω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν πρόκειται για τροποποίηση ούτε των επιχειρησιακών σχεδίων που δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν για να εφαρμοστεί το σύστημα, ούτε τροποποιείται το σύνολο του ε, χρηματοοικονομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας για κάθε χώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Δεν δίνονται περισσότερα κονδύλια, ούτε αμφισβητούνται σε καμία περίπτωση τα χρηματοοικονομικά πλαίσια τα οποία είναι διαθέσιμα για κάθε χώρα μέλος. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι εντός αυτού του χρηματοοικονομικού πλαισίου που δεν τροποποιείται, απλώς επιταχύνεται ε, η προκαταβολή που δίνεται από τα κοινοτικά κονδύλια. Επιταχύνονται λοιπόν η ε, διαδικασία πληρωμών ώστε να υπάρχει οικονομική ρευστότητα και να μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή τα προγράμματα τα οποία εξαρτώνται ε, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, εκτίμησε τις πρακτικές ε, πτυχές. Ε, υπολογίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ότι θα δοθούν 20 εκατομμύρια για τον προπολογισμό του 2012, δηλαδή μεταξύ των έξι χωρών μελών θα μπορούν να λάβουν ως προκαταβολή 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία χωρίς την παρούσα τροποποίηση του κανονισμού δεν μπορούσαν να λάβουν ως προκαταβολή. Έχουμε λοιπόν 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, μία ένεση κονδυλίων ώστε να μπορούν ε, να εφαρμόσουν καλύτερα τον ε, κανονισμό για το 2012. Ε, επίσης κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Έχουν συμφωνήσει στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη για αρκετά ζητήματα και το Κοινοβούλιο βεβαίως ε, είναι ενήμερο για τους συμβιβασμούς στους οποίους καταλήξαμε, αλλά εκρεμούν κάποια θέματα. να έχουμε ίσως δυνατότητα αναδρομικής ισχύω ώστε χώρες ε, όπως η Ουγγαρία που δεν εντάσσονται στο σύστημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας να μπορούν να υποφεληθούν του μηχανισμού για τους μήνες ε, στους οποίους ε, δεν είχαν ακόμα ενταχθεί. Επίσης, προτείνεται η εφαρμογή του μηχανισμού αυτού να μην είναι αυτόματη, αλλά να μπορεί η Ευρωπαϊκή εφαρμογή να έχει, ε, Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά στα κράτη-μέλη οι προτάσεις του Συμβουλίου, στις οποίες ε, κατέληξε και σε συμφωνία το Συμβούλιο, αλλά εξετάζει και τα υπόλοιπα ενδεχόμενα, όπως θα τα εξετάσει φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ο κανόνας ε, της αυτόματης αποδέσμευσης ε, εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι, εφαρμόζεται. Απλώς επιταχύνεται η διαδικασία. Δεν δίνεται περισσότερος χρόνος για την εφαρμογή των σχεδίων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φιγκερέιδα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, νομίζω πως ε, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε κάποιες ε, εξηγήσεις σε σχέση με τη θέση της. Θα ήθελα παρόλα αυτά να τονίσω τρία σημεία. Πρώτον, παρότι επιταχύνεται η διαδικασία, όπου και είναι θετικό, δηλαδή μια προσάυξηση της τάξης του 10% για κάθε πρόγραμμα. παρόλα αυτά δεν αυξάνεται το ύψος της χρηματοδότησης από πλευρές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια που προορίζονταν για ένα κράτος, δεν μπορεί να ε, καταβάλει επιπλέον πόσα η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Δηλαδή για προγράμματα που ήδη έχουν παρουσιαστεί υπάρχει μια αυτή η προσάυξη του 10%. Επιταχύνεται απλώ η διαδικασία. Μα είναι κρίμα. Διότι οι χώρες που είναι σε μια τέτοια κατάσταση αντιμετωπίζουν σοβαρές ε, δυσκολίες ε, ως προς την εθνική χρηματοδότηση πιστεύω πως θα έπρεπε να επανεξετάσει αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι για την προκειμένη περίπτωση, ενώ να το επανεξετάσει εν ώψη των μελλοντικών εξελίξεων, γιατί πιστεύω ότι οι δυσκολίες θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη για τα επόμενα χρόνια. Για του χρόνου, λοιπόν, καλό θα ήταν να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε, να επανεξετάσουμε το θέμα για να βελτιώσουμε το σύστημα. Γιατί αυτές οι χώρες, και εγώ από εκεί είμαι, το γνωρίζετε, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται αυξημένη χρηματοδότηση, αυξημένη στήριξη πέρα του 10%. Ε, και, μέσα, για κάποιες περιπτώσεις θα χρειαζόταν επανατροφοδότηση, αν θέλετε, του Εθνικού Κονδυλίου. Άλλη μια σημαντική πτυχή είναι η αναδρομική ισχύ. Νομίζω προβλέπεται εξ αρχής να αρχίζουν να ε, περιέρχονται αυτές οι χώρες σε μια κατάσταση οικονομικής αρρωγής, ας το πούμε έτσι. Ε, και νομίζω ότι ε, η Ουγγαρία ενδέχεται μόνο να βγει από αυτή την κατάσταση, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς τι είπατε για αυτό το σημείο. Δεν ήταν πολύ σαφές για μένα. Όπως είπατε, Πρόεδρε, ο εισηγητής εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέλευση των χωρών ΑΚΕ. Δεν υπάρχει, ε, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ε, πρόβλημα με την παρουσίαση της θέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά καλό θα ήταν ε, να μας υποβάλει τη θέση της για να... Εντάξει, μας είπατε ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές τροποποιήσεις, αλλά θα το ήθελα και γραπτό αν δεν σας κάνει κόπο. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις δύο ερωτήσεις που διατύπωσε η κύριε Το αναδρομικό στοιχείο εφαρμόζεται από τη στιγμή που η χώρα, όποια και αν είναι, όχι μόνο η Ουγγαρία, που εφαρμόζεται ο μηχανισμός. Αυτή στιγμή δηλαδή το κράτος μέλος ε, υποβλήθηκε στην ε, χρηματοοικονομική στήριξη. Αναφέρθηκα στην Ουγγαρία γιατί η Ουγγαρία είναι ειδική περίπτωση διότι δεν εντάσσεται στο μέσο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αλλά ε, μπορεί παρόλα αυτά να υποφεληθεί του μηχανισμού για την περίοδο στην οποία βρισκόταν στο χρηματοοικονομικό μηχανισμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ισχύει αναδρομικά μόνο για την Ουγγαρία, ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη από τη χρονική στιγμή στην οποία άρχισαν να λαμβάνουν χρηματοοικονομική στήριξη για τη μη τροποποίηση των ε, ταμείων, σας το επιβεβαιώνω, όντως αυτό που κάνουμε εμείς είναι απλώς ε, να επιταχύνουμε την ε, πληρωμή των κονδυλίων. Δεν αλλάζει ούτε το σχέδιο, ούτε το συνολικό ποσό το οποίο έχει καθοριστεί ότι θα λάβει κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Κάτι άλλο, κύριε Φιγκερέιδο, τίποτα άλλο. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Φιγκερέιδο, η οποία ανέλαβε να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρέμβασή της και προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Α, συγγνώμη, 28 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι τροπολογίες. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με το σημείο 7 και περνάμε στο σημείο 10. 11, συγγνώμη, ανταλλαγή απόψεων με τον Πασκάλ Σαβουρέ, Γενικό Διευθυντή της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλίας του ΒΙΚΟ. Έχετε το λόγο, καλώς ορίσατε και σας δίνουμε το λόγο. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή σας συνεδρίαση. Είμαι εκτελεστικός διευθυντής της ε, Νοσιακής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιέας του Βίγκο και θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα απολογισμό των εργασιών για το 2011 για την υπηρεσία. Ε, το ολοκληρώσαμε στις 23 Νοεμβρίου και θα ήθελα να παρουσιάσω και τις κατευθυντήριες γραμμές που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 18 Οκτωβρίου και παρουσίασε τις προτεραιότητες για το 2012 συγγνώμη, θα σας τις εκθέσω και ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το μέλλον της υπηρεσίας. Όπως γνωρίζετε, η υπηρεσία βασίζεται σε κοινά ε, προγράμματα ανάπτυξης πόρων, Joint Deployment Program, ε, υπάρχουν διάφορα, βλέπετε το ένα με το κόκκινο χρώμα στην παρουσίαση. Ο συντονισμός των εθνικών μέσων από την υπηρεσία οδήγησε σε 346, 346 ε, ελέγχους ε, στα σκάφη ε, και συνολικά ελέγχθηκαν 659 ε, τον αλλιευτικά. Συντονίζουμε λοιπόν τα εθνικά μέσα, αλλά όχι μόνο αυτό. Ε, ναυλώσαμε σκάφη από την υπηρεσία εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εφτάσαμε στις 240 ημέρες στη θάλασσα και συμπληρώθηκαν από 149 ημέρες ελέγχου και εκεί πρέπει να προσθέσετε όχι 68 ε, ημέρες ε, λειτουργίες, αλλά 68 ε, ημέρες ε, στη θάλασσα. Υπάρχουν θέματα τεκμηρίωσης, ε, παραδείγματος χάρη για τους δανέζικους γρήπους για την αλία τόνου. Υπάρχει το πρόβλημα των ε, ε, της ποιότητας ε, της ηλεκτρονικής καταγραφής από την κάμερα όταν περνάει το ψάρι από τη θάλασσα μέσα στη λεκάνη υποδοχής και το άλλο θέμα μας είναι το BCD το επωνομαζόμενο δηλαδή το η ηλεκτρονική καταχώρηση των αλλιευμάτων Υπάρχουν θέματα ε, συντήρηση σε σχέση, παραδείγματο χάρη, με την τήρηση του ελαχίστου μεγέθου του ερυθρού τόνου. Ε, επίσης σχέση με, ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα με το, ε, σε σχέση με το VMS, δηλαδή με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των σκαφών και άλλα ζητήματα που σχετίζονται γενικότερα με τις επιθεωρήσεις. Ε, στην τελευταία τακτική συνεδρίαση της ΣΥΤΑ της ΕΙΚΑΤ ε, που έλαβε χώρα στην ε, Κωνσταντινούπολη και τελείωσε συνεδρίαση το περασμένο Σάββατο, σε αυτή τη συνεδρίαση λοιπόν βελτιώθηκε κατά πολύ η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν δεχτήκαμε επικρίσεις όπως το παρελθόν και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συνολική συμμόρφωση ε, της ε, Επιτροπής σε σχέση με τα πρότυπα για τον ερυθρό τόνο έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό σχέση με το παρελθόν και νομίζω ότι αναγνωρίζεται και αυτό ε, στην ICAT. Ε, τώρα μια άλλη επιχείρηση σχετίζεται με την Βόρεια Θάλασσα ε, που ε, υποδιαιρείται σε διάφορα υποσύνολα. Έχουμε τις ε, σύντομε επιχειρήσεις, εννέα, το αριθμό στη Βόρεια Θάλασσα, και στην Δυτική Σκοτία δεν αναφέρεται εδώ γιατί αυτό εγγράφεται στα πλαίσιο ανάκαμψης του αποθέματος του γάδου ε, υπάρχει μια σχεδόν πάγια επιχείρηση που αρχίζει τον Ιανουάριο, πάει μέχρι τον Ιούνιο και μετά επαναλαμβάνεται στα τέλη του έτους και κινητοποιούμε μεγάλο αριθμό μέσων για αυτή. Βλέπετε ότι ε, στην επιχείρηση στη Βόρεια Θάλασσα έχουμε μια μεγάλη ε, ευελιξία διότι αναπτύσσουμε αυτή την έννοια των ε, σκαφών του βασικού ελέγχου, των συνδεδεμένων σκαφών, ούτω ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία όταν, χρειάζεται μια, όταν υπάρχει μια ad ανάγκη ελέγχου σε μια συγκεκριμένη ζώνη δηλαδή. Ε, τώρα το θέμα εντοπισμού θέσης, ε, στίγματος μάλλον μέσω δορυφόρου. Και στα πλαίσια αυτού του κοινού επιχειρησιακού προγράμματο υπάρχει διαρκή διαβούλευση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Οι επιθεωρήσεις ε, βασίζονται στην ανάλυση του κινδύνου και στη, σε μία πολύ ε, προηγμένη στοχοθέτηση η ε, συνεχώς ελέγχονται οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της εγκύτητα σε των υδάτων που όμως υπόκειται, εντάσσονται μάλλον σε διαφορετικές ε, επικράτειες. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, οι επιθεωρητές. Ή μάλλον ε, υπάρχει μεγάλη ενοποίηση, αν θέλετε, των εθνικών μέσων αυτών των χωρών και πιστεύω ότι πρέπει ε, να ε, προωθήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω το σύστημα, κυρίω στα πλαίσια των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ε, τα σχέδια επιθεώρηση για το μπακαλιάρο. Έχουμε δύο υποζώνες. Όπως βλέπετε, ο αριθμός των σκαφών που επιθεωρήσαμε στην επιχείρηση ε, φτάνει τα 544 ε, με 504 επιθεωρήσεις κατά την εκφόρτωση ε, και στη διακεκομένη επιχείρηση 418 σκάφη στο σύνολο 331 στην εκφόρτωση. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο αριθμός των παρατυπιών σχετίζονται με τις υποχρεώσεις αναφοράς. Δηλαδή, ε, σχετίζονται με ε, το αν αληθεύουν οι δηλώσεις ή με το αν υπάρχουν λάθη, σοβαρά σφάλματα ε, σε σχέση με τις ποσότητες που καταχωρούνται στο ημερόλογιο του πλοίου ή που δηλώνονται. Σε σχέση τώρα με το μέγεθος των δίχτυων, των ματιών των δίχτυων, πριν από λίγες εβδομάδες πιάσαμε ένα σκάφος με ένα σύστημα που ονομάζουμε blinders στα αγγλικά, σωσέτ στα γαλλικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουν ε, ακόμη προβλήματα διότι υπάρχουν δίχτυα που δεν είναι καθόλου συμβατά με τα μέτρα ε, διατήρησης. Υπήρξαν και προβλήματα με τις άδειες 27 ε, παραβιάσεις με έγγραφα επιπρόσθετα που συνδέονται με την διαχείριση του αποθέματος του γάδου και σχετίζονται με τις αλληλευτικές ε, προσπάθειες. Ε, κατά τα λοιπά, αυτό το κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα μας επέτρεψε να εντοπίσουμε 139 σκάφη που είχαν διαπράξει τουλάχιστον μία ε, παρατυπία με, σε σχέση με 1.300 περίπου σκάφη που επιθεωρήσαμε στο σύνολο και 1500 περίπου που ελέγξαμε ε, στην ε, εκφόρτωση. Ε, αυτά για το γάδο. Για το σολομό δεν εντάσσεται ακόμη στο κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα, αλλά είναι θέμα χρόνου. 393 πλοία επιθεωρήσαμε στο σύνολο είχαμε 109 μέρες επιχειρήσεων ε, στο χρόνο, αλλά τα προβλήματα σχετίζονταν περισσότερο με την πρώτερη άδεια, ήταν ζητήματα των ειδικών αλλιευτικών αδειών, γιατί το είδος αυτών των παραβιάσεων φτάνει στις 29, όπως βλέπουμε. Ε, άλλα προβλήματα σχετίζονταν με τις ε, δηλώσεις των ποσοτήτων και αυτό είναι πιο ανησυχητικό διότι φτάσαμε 18 παραβάσεις. Ε, θα ήθελα επίσης ε, να σημειώσω ότι η συνεργασία με τη Ρωσία ξεκίνησε φέτος, ε, κυρίως το Σεπτέμβριο του 2011, όπου ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης μετήχε σε ένα εργαστήρι για την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα. Ήταν εξαιρετικά θετική αυτή η εμπειρία. Ε, τώρα το κοινό πρόγραμμα για τα δυτικά ύδατα είναι ένα νέο σύστημα που εισήχθη φέτος ε, στις 5 Σεπτεμβρίου 2011 άρχισε να τρέχει αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα ε, που καλύπτει προφανώς σε διάφορα είδη, καλύπτει όλα τα πελαγικά είδη με την εξαίρεση ε, προφανώς των ειδών ε, που, για τα οποία είναι αρμόδια η ΑΕΚΑΤ. Ε, έχουμε τις, το γάβρο, τη ρέγγα και άλλα είδη. Είναι λεπτό το ζήτημα, διότι σίγουρα γνωρίζετε το πρόβλημα για το σκουμπρί σε σχέση με τις αυτόνομες ποσοστώσεις που πήραν εντελώ μονομερός ε, κάποια παράκτια κράτη της Βαλτικής ε, για αυτό το είδος. 32 ε, σκάφη επιθεωρήσαμε στη θάλασσα και 194 στην εκφόρτωση. Το θέμα, τα, οι παρατυπίες μάλλον σχετίζονται και πάλι εδώ με τις δηλώσεις. Πρόκειται για ένα κοινό ε, επιχειρησιακό πρόγραμμα που παρουσιάζει, όπω σα είπα, δύο ιδιαιτερότητε. Ε, πρώτον, ε, ήδη αναφέρθηκα στο ότι καλύπτει πληθώρα ειδών και δεύτερον, είναι πάγιο. Πρόκειται για μόνιμη δομή ω προ το επιχειρησιακό σκέλο, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη. Euh, euh, Άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει διάφορα είδη είναι αυτό που καλύπτει την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή στη σχέση στα πλαίσια των διεθνών δεσμεύσεων ε, βόρειο, δυτικός και βόρειο Ατλαντι, ανατολικός Ατλαντικός ε, ΝΑΦΟ και ΝΕΑΦΚ δηλαδή ε, επιθεωρήσαμε 32 σκάφη ε, στη ζώνη ΝΑΦΟ και 112 στη θάλασσα για τη ζώνη που ελέγχει η ΝΕΑΦΚ. Ε, οι παρατυπίες εν γέννη σχετίζονται ε, με το θέμα των αδειών, των αλληλευτικών δικαιωμάτων, καθώς και με την ε, την ε, δήλωση των ε, ειδών που αλλιεύονται. Ε, υπάρχουν άλλες παρατυπίες που διαπιστώσαμε στις κοινές επιθεωρήσεις που κάναμε με τον Καναδά. Ε, και πάλι εδώ οι επιθεωρητές έπαιξαν τον ρόλο των ε, επιθεωρητών της Ένωσης. Επίσης ε, κάναμε και ένα κοινό σεμινάριο. οι Καναδοί που είχαν αναλάβει ε, τις επιθεωρήσεις, ε, πρόσωπός τους μάλλον θα έρθει σε μια συνεδρίαση που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στο Βίγκο. Έχουμε πάρα πολύ καλές ε, σχέσεις και θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία, αυτή την εμπιστοσύνη που υπάρχει. Όπως ξέρετε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασιστικό ρόλο ε, διότι μπορέσαμε να αναβλώσουμε φέτος ένα σκάφος ε, για τις επιθεωρήσεις ε, με κόστος 4 εκατομμύρια για να ικανοποιήσουμε και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τηλεγραφικά σας πω ότι χρησιμοποιήσαμε τρεις μήνες για τον ερυθρό τόνο και τέσσερις για τις ζώνες ΝΑΦΟ και ΝΕΑΦΚΑ. Ε, βλέπετε πως η δραστηριότητα ε, ε, για αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανήλθε σε 79 μέρες και στελεχώθηκε και από επιθεωρητές τρίτων χωρών, από την Τουρκία παραδείγματος χάρη, 91 συναλλιευτικά επιθεωρήθηκαν και ανακαλύψαμε παρατυπίες μετά από αυτές τις επιθεωρήσεις. Στις ζώνες που ελέγχει η ΝΑΦΟ και η ΝΕΑΦΚΑ ε, Έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό ημερών εν πλώ, αλλά ε, ο αριθμός των επιθεωρηθέντων πλοίων είναι χαμηλότερος, ε, δεδομένης και της Ευρύτητα των υδάτων και τη στενότητα των μέσων που έχουμε για να καλύψουμε αυτές τις ε, μεγάλες ζώνες. Ε, για το σκάφος αυτό που ναυλώσαμε βλέπουμε διάφορα θετικά σημεία διότι πρώτον ε, καταδεικνύουμε πόσο ισχυρή είναι η διεθνής δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σκάφος αυτό, όπως βλέπετε, είναι Ισλανδικό. Ε, προαγάγει την ανταλλαγή απόψεων τη συνεργασία ανάμεσα στους επιθεωρητές Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους επιθεωρητές των τρίτων χωρών με στόχο την εναρμόνιση των ε, πρακτικών και στα πλαίσια της ΕΚΑΤ να υλοποιήσει το Διεθνές Πρόγραμμα Ελέγχου του Ερυθρού Τόνου της ΑΕΚΑΤ ε, και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο το σκάφος αυτό για τους εν λόγω ελέγχους. Ήδη αυτή είναι η επιχειρησιακή δραστηριότητα της υπηρεσίας, έτσι μπορούμε να την περιγράψουμε μέχρι ε, στιγμή στα πλαίσια, είπαμε, των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ε, τώρα, σε σχέση με το πρόγραμμα εργασιών ε, το, της υπηρεσίας για το 2011, προφανώς φέρουμε σοβαρή ευθύνη στα πλαίσια του ε, συντονισμού τη ε, της δράσης των κρατών μελών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στα κράτη-μέλη δηλαδή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την καταπολέμηση της λαθρέας επάνωσης και αναρχιθαλίας. Η συμμετοχή της υπηρεσίας έγκυται στην ε, ε, υλικοτεχνική υποστήριξη κατά τις επιθεωρήσεις σε τρίτες χώρες, ε, στη Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Παπουασία, Νέα, Παπουασία, Νέα Γουινέα. ούτω ώστε οι χώρες αυτές που εξάγουν ε, προϊόντα προς την εσωτερική αγορά να συμμορφώνονται με τις απαιτήσει υποχρεώσει περί διατήρηση των αποθεμάτων. Οργανώσαμε επίσης εργαστήρια για να γίνει ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στους επιθεωρητές. και για να ε, παρουσιαστούν οι βέλτιστες ε, πρακτικές, ούτως ώστε να ισχύουν ε, ίσοι όροι για όλους ε, και κυρίως ομοιόμορφοι. Οργανώσαμε την περασμένη εβδομάδα ένα άλλο εργαστηρί, παρουσία εκπροσώπων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, στα πλαίσια ε, της ε, σύμβασης πονήμε και συγκεκριμένα το άρθρο 188 σε σχέση με τη δραστηριότητα των αλλιέων και ε, πραγματικά υπάρχουν λυπηροί όροι εργασία εν πλώ και αυτό ε, καταδεικνύει ότι παραβιάζονται οι κανονισμοί γιατί δεν, γιατί δεν υπάρχει ε, παρκής ανταλλαγή ε, απόψεων. Πέραν αυτού η υπηρεσία για να εξυπηρετήσει τα κράτη-μέλη και για να προσφέρει αυτή την υγροτεχνική στήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θέλει να αναπτύξει τα μέσα της και έτσι μία από τις δράσεις μας ήταν να κάνουμε μία απογραφή των συστημάτων πληροφορικής και ενημέρωσης των ε, κρατών μελών με στόχο την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τους ε, ελέγχους ε, για... και με στόχο τον προσδιορισμό των βελτίστων πρακτικών ούτως ώστε να διαδοθούν. Ως προς την κατάρτιση και την ενημέρωση ένα εγχειρίδιο εκπονήθηκε ε, που προορίζεται ε, στους εκπαιδευτές των επιθεωρητών και τους ίδιους τους επιθεωρητές ε, για την επιθεώρηση, θαλάσσια επιθεώρηση, η υπηρεσία εντάσσεται, συμμετέχει μάλλον στην πρωτοβουλία ΣΥΣ συνεργαζόμαστε με τη Frontex και την ΕΣΑ στα πλαίσια μιας ε, κοινή ε, ομάδας εμπειρογνωμόνων. Η πρώτη δοκιμή ανταλλαγής ε, δεδομένων για εικόνες που σχετίζονται με την θαλάσσια παρακολούθηση οργανώνεται και Προφανέστατα σε αυτό εντάσσεται και η ναύλωση του σκάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ελέγχους που ήδη ανέφερα. Ο προϋπολογισμός βασίζεται σε τρία τμήματα, διοικητικές ε, δαπάνες που για το 2012 προβλέπεται στα 6,58 ε, εκατομμύρια. Οι λειτουργικές δαπάνες θα ανέλθουν για το 2012 σε 1,73 ε, και άρα υπάρχει μια ένα συνολικός προϋπολογισμός ε, της τάξης ε, των 9,31 εκατομμυρίων. Ε, ξέρουμε όμως ότι θα μειωθεί τελικά ο συνολικό προπολογισμό κατά 1%. Το μάθαμε πριν από λίγε μέρες. Θα πρέπει λοιπόν ε, λόγω των δημοσιονομικών ε, περιορισμών ε, να περιοριστούμε κι εμείς και θα αφαιρεθεί αυτό το 1%. Πάντως, ο προϋπολογισμός αυτό προβλέπεται από την αντίστοιχη οδηγία, ο προπολογισμό για το 2012 θα απορροφηθεί κατά 98% όπως εξάλλου και το 2010. Για να γυρίσω πίσω, ο προϋπολογισμός του 2011 συμπεριλαμβάνει και τη χρηματοδότηση ε, της ναύλωσης αυτού του ε, σκάφους και το 2012 ως προς ε, τις επιστώσεις πληρωμών υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ διότι έχουμε πιστώσεις πληρωμών ενός εκατομμυρίου που θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία αυτού του σκάφους ε, λίγη στις 31 Μαρτίου αυτή η πίστοση και γι' αυτό υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πιστώσεις ανάληψης υποχρέωσεων και τις πιστώσεις πληρωμών ενός εκατομμυρίου. Nous sommes donc en de για την, ε, για την απορρόφηση των κομιλίων τα είπα ήδη, δεν επιμένω τώρα ως προς την κατανομή του προσωπικού, ως προς τις δραστηριότητες της υπηρεσίας ε, βλέπετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι σχετίζεται με τις επιχειρησιακές δαπάνες, ε, καταπολέμηση δηλαδή τις παράνομες λαθρέες και ανερξελίας και τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα. Ε, το 1 τέταρτο αντιστοιχεί στην ε, διαχείριση, τη διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό να έχουμε εργαλεία λογισμικού που θα βοηθήσουν την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ο επιχειρησιακός ε, συντονισμός ε, αντιστοιχεί στο 72% το 13%, το 9% του προϋπολογισμού χρησιμοποιείται ε, για τα διοικητικά για τη χρηματοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2011 ε, αριθμούσε το προσωπικό μας 62 άτομα και 4 αποσπασμένοι εθνικοί απορρογνώμονες. Ε, το 2012 θα μπορούσε να αυξηθεί το προσωπικό κατά έναν υπάλληλο αλλά, αλλά ε, λόγω των ε, περιορισμών ε, δεν είναι σίγουρο αν θα προσληφθεί αυτός ο υπάλληλο. Αυτά εντάχει για το 2011, δεν έχει βεβαίως λήξει. Θα ήθελα όμως τώρα να αφήσουμε το 2011 και να μιλήσουμε για τον προγραμματισμό του 2012 ή και των επόμενων ετών. Ε, ως προς τα βασικά ε, ε, στοιχεία του κεντρικού κανονισμού του 768 της 26 Απριλίου του 2005 η υπηρεσία έχει ως εντολή να συμβάλλει ε, στην βιώσιμη διαχείριση των πόρων στον συντονισμό των εθνικών πόρων και στο συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι να υλοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο ο πυρήνας ε, της ε, ε, κοινής αλληλευτικής πολιτικής, δηλαδή η τήρηση των αλληλευτικών αδειών, των αλληλευτικών προσπαθειών, των, προσ... ποσοστώσεων για τις αλληλευτικές προσπάθειες και των... Και Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε ισότιμη μεταχείριση, ομοιόμορφου όρου που θα ισχύουν για όλου του επαγγελματίες του κλάδου. Να μην υπάρξουν δηλαδή διαφοροποίησεις, τρευλώσεις ε, λόγω διαφορετικής μεταχείρισης. Ε, αυτή η διάσταση είναι ακόμη πιο επίκαιρη σήμερα σε σχέση με την ίδρυση της υπηρεσίας το 2005 λόγω της κρίσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα μέσα που διαθέτουμε, να μην κατασπαταλούμε δηλαδή τα χρήματα του προπολογισμού ούτε και τους ανθρώπινους πόρους. Για το 2012 είναι σημαντικό να ε, επικεντρωθεί στην εντολή της η υπηρεσία, να προσφέρει στην υλοποίηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μίλησα για την ε, συμμόρφωση με τα πρότυπα του κανονισμού. Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με τη χρηματοδότηση και η τρίτη με ε, την ομοιομορφοποίηση των όρων που ισχύουν επί τόπου. Ως προς την ε, διαχείριση και υλοποίηση των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι σαφές ότι οι δείκτες επιδόσεων, η οικονομική αποτελεσματικότητα και η ανάλυση του κινδύνου είναι τρεις συνιστώσεις που θα πρέπει να ε, αναδειχθούν σε ε, βασικές αυτές αρχές της υπηρεσίας θα πρέπει η υπηρεσία να προσφέρει στήριξη όχι μόνο προς ε, τα κράτη-μέλη, όχι μόνο ως προς τη χρησιμοποίηση του συνόλου των πόρων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να επικουρεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη η διακυβέρνηση η διαχείριση ε, μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθεί ε, σε στρατηγικού χαρακτήρα σχέδια ώστε να επαναπροσδιοριστεί ίσως ε, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε ε, νομικά και επιχειρησιακά μέσα, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και τους ε, δείκτες επιδόσεων καθώς και η ιεράρχη των προτεραιοτήτων, ούτως ώστε οι στρατηγικές κατευθύνσεις που δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο να παρακολουθούνται, να βελτιώνονται αν χρειάζεται και να εφαρμόζονται στην πράξη. Για το 2012 Ε, καλή την υπηρεσία να εφαρμόσει το πρόγραμμα εργασιών ε, που ε, συζήτησε και ενέκρινε 18 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο και πάλι εδώ επιδιώκουμε να προσφέρουμε τις πλέον αποτελεσματικές υπηρεσίες ε, για, με στόχο την ε, ορθή εφαρμογή της κοινής ελευτικής πολιτικής ε, και θα επικεντρωθούμε σε δύο βασικές δραστηριότητες, επιχειρησιακές, επιχειρησιακού χαρακτήρα, δηλαδή κοινά επιχειρησιακά προγράμματα και δεύτερον ανάπτυξη των ικανοτήτων κυρίως ε, ως προς την κατάρτιση τα εγχειρίδια και η υποστήριξη των επιχειρήσεών μας, δηλαδή ανάλυση κινδύνου, ε, παροχή ε, δεδομένων. Ο απότερο στόχος είναι να υπάρξει καλύτερη γνώση ως προς την κατάσταση που επικράτει μέσω συλλογής ε, στοιχείων που κοινοποιούν τα κράτη-μέλη για τα αλλιεύματα του εθνικού του στόλου αυτή η συλλογή στοιχείων έχει κέριο κεντρικό ρόλο στη δράση της ε, υπηρεσίας μας. Ε, βλέποντας αυτό το πρόγραμμα για εργασίες για το 2012, ε, εκ πρώτης όψης δεν διαπιστώνουμε κάποιες σοβαρές αλλαγές σε σχέση με το 2011. Με όλα τα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε κάποιες δράσεις αρρωγή προς την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και στα πλαίσια της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ε, στη Μεσόγειο, συγκεκριμένα χώρες της Αραβικής Άνοιξης όπως λέμε, με την Τουρκία, την Κροατία. Ενάν, νέο δημοσιονομικό δελτίο και δελτίο καθηκόντων ε, καταρτίστηκε για τα δυτικά ύδατα. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο ε, που ε, συζητούμε εδώ και μήνες. Δηλαδή, από την περιφερειακή διάσταση μετακινόμαστε προς μια προσέγγιση που είναι συνάρτηση των ειδών. Σας μίλησα για την Βόρεια Θάλασσα, ε, για την ε, Μεσόγειο, για τον Ατλαντικό, για τον Ερυθροτόνο, ε, για 63 διαφορετικά είδη. Και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούν να έχουν αυτή την περιφερειακή διάσταση, ούτω ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση των, των θεμάτων διατήρηση του αποθέματος σε περιφερειακό επίπεδο να υπάρχει ενοποίηση των προσπαθειών Στα πλαίσια αυτών των προτεραιοτήτων δεν πρόκειται να σημειωθούν σημαντικές διαφορές ως προς την λαθρέα παρανομική αναρχιαλία. Θα συνεχίσει τη δράση της η υπηρεσία και θα συνεχίσει να εξετάζει ε, μελλοντικές δράσεις στον τομέα αυτό. Ε, έγινε στο Ζοπότ στις 25-26 Ιουλίου φέτος μία συνεδρίαση στα πλαίσια της Πολωνικής Προεδρίας ε, με στόχο να εξετάσουμε ε, νέες δυνατές δράσεις για την καταπολέμηση της παράνομης λαθρείας και ανεξαλίας. Πάλι για το 2012 το δελτίο που σχετίζεται με τη θαλάσσια επιθεώρηση επιφέραμε κάποιες αλλαγές ώστε ε, να φανεί ποιος είναι ο ρόλος της ε, υπηρεσίας στα πλαίσια της ε, ενιαίας θαλάσσιας πολιτικής χρησιμοποιώντας μέσα που παλιά χρησιμοποιούσε η ΕΜΣΑ ή ο Frontex στον τομέα της ε, κατά πολέμησης της λαθρέας παράνομης αναρχισαλίας ε, και στα πλαίσια των επιθεωρήσεων επίσης. Ε, θέλουμε να έχουμε διάφορα στρώματα ενημέρωσης να χρησιμοποιούμε δεδομένα VMS παραδείγματος χάρη ή δεδομένα ES ή δεδομένα από παρακολούθηση που γίνεται μέσω δορυφόρου διασταυρώνοντας τις εικόνες δορυφόρου έχουμε ε, στοιχεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ανεξαρτήτως ε, δράσης ε, το των σκαφών. Έτσι μπορούμε να έχουμε ομοιόμορφη ενημέρωση ε, Βεβαίω, στα πλαίσια που τα κράτη-μέλη θα δεχνούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα νέα έντυπα. Η συνδρομή προ την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, για την συνεργασία με τις τρίτες χώρες, κυρίως ως προς τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης ε, δεδομένων και ενημέρωσης, το URS συγκεκριμένα, αλλά και το FISNET όπως ονομάζεται, ε, όπου αναγράφονται όλες ε, οι πληροφορίες σε σχέση με τις επιθεωρήσεις που γίνονται στα πλαίσια των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων με στόχο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ε, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας μίλησα ήδη για την νέα θαλάσσια προσέγγιση και κυρίως για την πρωτοβουλία ΣΥΣ που μαζί με τη ε, αν θέλετε μαζί με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ ε, η υπηρεσία μας ε, είναι ο αλληλευτικός εμπειρογνώμονας γιατί πρόκειται για δεδομένα που είναι κέρια σημασία για να συμπληρώσουμε τη δράση των μέσων μας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Σας μίλησα για την χρησιμοποίηση νέων πόρων για νέες αγορές, αλλά ε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο για το 2012 λόγω των περιορισμών που προανέφερα. Θα πρέπει να εξακριβώσουμε αν ε, ε, χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους και να προσπαθήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τη δράση της υπηρεσίας. Παραδείγματος χάρη πιο αντίκτυπο είχαμε ως προς την βιωσιμότητα της διαχείρισης κάποιων αποθεμάτων. Σας είπα επίσης να εργαστούμε περαιτέρω για την ελεγξιμότητα, ζητώ συγγνώμη για αυτή τη λέξη, την ελεγξιμότητα λοιπόν ε, της, ε, των πόρων, της χρήσης των πόρων. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η έλεγχη Πρέπει να γνωρίζουμε ε, ε, τα μέσα των κρατών μελών ε, ως προς τις ζώνες, τον αριθμό ημερών, των πόρων τους, το κόστος που συνεπάγεται κάθε πρόγραμμα για το κράτος μέλος και να προσπαθήσουμε να σε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρούμε νέα μέσα για να ενισχύσουμε την προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα της δράσης μας. Η ανάγκη ελέγχων, η έλεγχη μάλλον δεν είναι η μόνη ε, παράμετρος ε, για ε, υπέρ της ε, βιωσιμότητας ε, οι δράσεις καταστολής που αναλαμβάνει η υπηρεσία μας επίσης συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας. Το 2012 θα συνεχίσουμε υπό τον έλεγχο βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαθέτει το μονοπόλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Έχουν αρχίσει συζητήσει για ένα πρόγραμμα, ένα ειδικό πρόγραμμα ε, επιθεωρήσεων και ελεγχών είναι ένα νομικό εργαλείο που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού μπορέσουν να υλοποιηθούν κοινά επιχειρησιακά προγράμματα ως προς την περιφερειακή ε, διάσταση είναι σαφές ότι ότι ε, εφόσον θέλουμε να καλύψουμε πολλά είδη πλέον, ε, ε, θα είναι πολύ πιο περίπλοκα τα ζητήματα σε σχέση με το παρελθόν. Για την περιφερειακή διάσταση, τρει ζώνε όμω απασχολούν όλου ιδιαίτερω. Η Βόρεια Θάλασσα, η Βαλτική και τα δυτικά Ήδατα. Ίσως υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις ίσως σημασίας, αλλά αυτό πάντως το στοιχείο έχει μεγάλη σημασία ως προς την μελλοντική διαχείριση των πόρων. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και μέσων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, όπως σας έλεγα προηγουμένως, αυτή είναι η επόμενη διαφάνεια. Ε, προσπαθούμε να να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση για την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και άναρχης ε, αλίας. Θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ε, και το 2012 και θα το εξετάσουμε, αλλά και πέραν αυτού. η υπηρεσία μας ε, θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την αναθεωρημένη κοινή αλληλευτική πολιτική. Αυτό το discard ban, η απαγόρευση των απορρίψεων, είναι ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι προφανές πως η υπηρεσία μας ε, θα αρχίσει να διοχετεύει πόρους σε αυτό το τόσο περίπλοκο ζήτημα κάτω την ετοιμότητα των κρατών μελών. Πέραν αυτού, ε, προβλέπεται και μια εξωτερική επιθεώρηση της υπηρεσίας μας σε βάση του κανονισμού. Τώρα διεξάγεται αυτή η εξωτερική επιθεώρηση. Η, η έκθεση... Ε, θα ε, ε, ε, εκπονηθεί σε 6 Φεβρουαρίου του 2012 από δύο εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που θα αξιολογήσουν τη δράση της υπηρεσίας στα πλαίσια στα πλαίσια τη, μιας πρότασης αναθεώρησης του κανονισμού δημιουργίας ή ίδρυσης του, της ίδιας της υπηρεσίας, αλλά δεν θα επεκταθώ σε αυτό γιατί είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ως προς τη μετεξέλιξη του νομικού πεδίου δράσης της υπηρεσίας νομίζω ότι το θέμα της ε, διάρκεια και το θέμα των θαλασσίων επιθεωρήσεων για την καταπολέμηση τη λαθρέα άνερχη και παράνομη αλίας θα είναι δύο πολύ βασικά στοιχεία στα πλαίσια αυτή τη του κανονισμού. Για την περίοδο μέχρι το 2020 είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη δράση θα πρέπει να απηχείται, να καταγράφεται στον προπολογισμό. Βλέπετε ότι ε, εξαντλούμε τα διαθέσιμα στην υπηρεσία μέσα δεν ε, διαθέτουμε πρόσθετους πόρους, εξού και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για το 2012, διότι δεν έχουμε πρόσθετους πόρους ούτε και επιπρόσθετο προσωπικό. Και ε, δεδομένης κατάσταση είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα. le fait que le, rapport sera disponible en sera Η έκθεση αξιολόγηση σας είπα θα είναι έτοιμη το 2012, θα συζητηθεί αυτή η έκθεση σε ένα ε, φόρουμ, σε ένα σεμινάριο που θα συνδυαστεί με την ε, σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου το Μάρτιο και τότε θα μπορέσει το Διοικητικό Συμβουλίο να λάβει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης. Εν κατακλείδη, ε, θέλω να τελειώσω με μια πρόσκληση είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στην σχέση με τα τρία θεσμικά όργανα. Με τα κράτη-μέλη έχουμε ε, μόνιμες πάγιες σχέσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και τον ε, Ιούνιο το 2010, θα χαρούμε όλος ιδιαιτέρως και εγώ και οι συναδελφοί μου να σας υποδεχτούμε στην υπηρεσία μας ε, όποια στιγμή, ε, στην υπηρεσία μας όποια στιγμή ε, κρίνετε ότι θέλετε να μας επισκεφτείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. una ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαβουρέ, για την ε, πολύ εκτεταμένη και δεξιοδικότατη παρουσίαση των σχεδίων της υπηρεσίας ελέγχου. Έχει ζητήσει καταρχάς το λόγο ο κύριος Ντέιβις. Thank you, Chairman, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Σαβουρέ για την παρουσίασή του. Επανέρχομαι στα στατιστικά στοιχεία για τις επεσορίσεις των σκαφών. Εντάξει. Ένα λεπτό. Okay, thank you. Um, we've all done that. Um... Ευχαριστώ λοιπόν τον εκτελεστικό διευθυντή για την παρουσίαση του. Αν μπορούμε να επανέλθουμε στα πρώτα στατιστικά στοιχεία για τις επιστολές των σκαφών. Αναρωτιέμαι αν μπορούσατε να μας ε, δώσετε μια καλύτερη εικόνα της όλης διαδικασίας από τα στεγνά στατιστικά στοιχεία. Καταρχάς, τι είδους συνεργασία λαμβάνεται από τους ε, όταν ε, ε, καταφθάνουν οι επιθεωρητές. Πώς τους υποδέχονται, τους καλωσορίζουν ή τους τέλος πάντων πώς τους δέχονται, πώς γίνονται αποδεκτοί οι επιθεωρητές. Δεύτερον, αναφέρεται στις, ε, στα λάθη τα οποία επισημαίνονται στις ε, εκθέσεις, στις αναφορές ε, τι, τι εννοείται με λάση, εννοείται παραπτώ, παρα, παρατυπίες απλές ε, ή παραβιάσεις, αδικήματα δηλαδή, <coughs> λάθη τα οποία μπορούν να θεωρηθούν αδικήματα, σοβαρά. Και τρίτον, όπου σημειώνονται αυτές τις παρατυπίες, αυτά τα λάθη, ε, τι διαδικασία ακολουθείτε, τι γίνεται μετά, αρχίζεται δικαστική διαδικασία, επιβάλλεται κυρώσεις, τι γίνεται μετά. Ευχαριστώ. Κυρία Λοβίν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Σαβούρα για την παρουσίασή σας. Έχω μερικές ερωτήσεις και μια παρατήρηση. Σε αυτή την επιτροπή εμείς δεν υπερψηφίσαμε την εξαιρετική, την επιπλέον γραμμή του Κοινοβουλίου για την ε, μίσθωση των ε, σκαφών επιθεώρησης και ελέγχου των ελεγκτικών σκαφών, ε, το οποίο ήταν μια λυπηρή μέρα και όχι καλή μέρα για την Επιτροπή μας. Τώρα, από τα στατιστικά στοιχεία που μας δείξατε, φαίνεται ότι οι περισσότερες παρατυπίες επισημάνθηκαν από τις επιθεωρήσεις που έγιναν εν πλώ στη θάλασσα. Πολύ περισσότερες από τις ε, παρατυπίες ή τα παραπτώματα που σημειώθηκαν στην ε, ξηρά. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η προσωπική σας άποψη ε, για τις επιπτώσεις του θαλασσίου ελέγχου εάν ε, η υπηρεσία σας δεν μπορέσει να μισθώσει ένα τέτοιο σκάφος για να εκτελέσει αυτές τις, αυτούς τους ελέγχους. Είδα επίσης από τα στοιχεία του προγράμματος του 2012 και τις ε, συντονιστικές ε, εκστρατείες, ε, συντονιστικά προγράμματα που θα κάνετε, ότι αναφέρονται στη Βόρειο Θάλασσα και όχι στη Βαλτική λοιπά και όχι στη Μεσόγειο. Θα ήθελε λοιπόν να σας ρωτήσω, θα συνεχίσετε με αυτούς τους ελέγχους στη Μεσόγειο ή όχι. Και τελευταία ερώτηση. Μόλις πληροφορήθηκα ε, της πρόοδους της τεχνολογίας που έχουν γίνει όσον αφορά τα μαύρα κουτιά, την ανάπτυξη μαύρων κουτιών ε, στα αλλιευτικά σκάφη όπως αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη. Το, μου φαίνεται ότι αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν θα θέλετε να ελέγξετε ε, τι ενέργειες έχει κάνει το λευτικό σκάφος και αν συμφωνεί με τις καταχωρήσεις στο βιβλίο κλπ. Ε, γύρω στα 500 ευρώ νομίζω κοστίζει η εγκατάστασή του δεν είναι και ακριβό το ποσό αυτό, δεν είναι πολύ και πιστεύω ότι θα είναι λίγαν αποτελεσματικό. Και τρίτον, χρησιμοποιείται ανάλυση DNA όταν, όταν κάνετε, σημειώνετε παρατυπίες στα λιεύματα ευχαριστώ. Euh, ε, θέλω να συμφωνήσω με την ερώτηση της κυρίας Λοβίν και να προσθέσω κι άλλες. Λοιπόν, πρώτα για τον ερυθρό τόνο. Είναι το πρώτο ζήτημα που σχολιάσατε. Έχω ε, μια αμφιβολία, ε, το ανέφερα χθε στην κυρία Δαμανάκη, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, που συζητήσαμε και στην Κωνσταντινούπολη για αυτά τα ευρωπαϊκά σκάφη που ε, αλείβαν στα ύδατα της ε, Λιβύης. Είναι διπλό το πρόβλημα. Ποιος είναι ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αρχίσει μια έρευνα τέτοιων περιπτώσεων ε, μετά από ε, σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας. Δηλαδή, χάρη στην υπηρεσία έχουμε το στίγμα ε, μέσω VMS για όλα τα σκάφη. Οπότε, ρωτώ, ποιος είναι ο μηχανισμός που έχει η υπηρεσία για να ενημερώνει και μετά για να αποδεικνύει ποιο σκάφος είναι εκεί που είναι και τι κάνει. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην ΑΕΚΑΤΕ θεωρείται ότι η υπηρεσία ε, λειτουργεί ε, ικανοποιητικά, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν κάποιες πτυχές που επιδέχονται σοβαρές βελτιώσεις. Δεύτερον, για τον ερυθρό πάλι, 79 ημέρες επιθεώρησης μας είπατε, με 16 επιθεωρητές και ε, επισκεφθήκατε 91 σκάφη. Πολύ απλό ερώτημα. Αρκεί. Αρκεί αυτό. Έχουμε αρκετά μέσα για να ελέγξουμε ολόκληρη την αλία του ερυθρού τόνου δεδομένη της ευρύτητας ε, των ζωνών ε, αλίευσης ε, και σε σχέση με τα προγράμματα ανάκαμψης που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη ερώτηση είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος, ε, θα μου πείτε αν έχω δίκιο ή όχι, ε, αλλά ε, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να έχουμε μια υπηρεσία που την ελέγχουν τα κράτη-μέλη, ενώ το αντίστροφο έπρεπε να συμβαίνει. η υπηρεσία έπρεπε να ελέγχει τα κράτη-μέλη. Εγώ διαπιστώνω ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό και οφείλουμε να το ρυθμίσουμε. Δηλαδή, το θέμα της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας και η δυνατότητα δράσης της υπηρεσίας και ελέγχου των κρατών μελών. Ε, συμφωνείτε Χρειάζεστε ε, μεγαλύτερη ανεξαρτησία για να ε, λειτουργήσετε ικανοποιητικά και δεδομένης της τωρινής κατάστασης δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα η υπηρεσία να δράσει ανεξάρτητα από τις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών και είναι κατάλληλη, πρόσφορη η κατάσταση τώρα για να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Παρακαλώ. Κύριο Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διευθυντή της Υπηρεσίας για την αναλυτικότατη παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση της ε, αλληλευτικής πολιτικής της Ένωσης. Θα ήθελα να θέσω τέσσερις ερωτήσεις. Πρώτον, με την πείρα σας αυτά τα χρόνια στη λειτουργία της υπηρεσίας, Θεωρείτε ότι προχωρήσαμε σε θέματα συνεργασίας και συμμόρφωσης από πλευράς κρατών μελών. Δεύτερον, για τους ελέγχους γίνονται επιθεωρήσεις ε, επί θαλάσσης και ξηράς. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω και στους επίγειους ελέγχους, διότι είναι και αυτή εξίσου σημαντική. Τρίτη ερώτηση, για τις τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπειρία από τη ε, λειτουργία της υπηρεσίας, θα μπορούσε ίσως να ήταν ενδιαφέρον να συνεργαστεί με χώρες τις οποίες ε, υπάρχουν ε, συμφωνίες αλληλευτικής σύμπραξης, υπάρχουν σχετικές προβλέψεις. Και τέλος, με την παρούσα δομή της υπηρεσίας, θα μπορούσε η υπηρεσία να αναλάβει κάποιες από τις ευθύνες οι οποίες απορρέουν από τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής για να ενισχυθεί το έργο τη. Η Πρόεδρος δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Θα ήθελα να θέσω και εγώ λοιπόν μια ερώτηση. Αυτό που θα ήθελα να μου πείτε είναι κατά πόσον στο μέλλον θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε και να διευρύνουμε κάποιες πτυχές της εργασίας της υπηρεσίας. Από ό,τι βλέπω, αυτή εξ αρχής η υπηρεσία έχει επικεντρωθεί σε τρεις ε, περιφερειακές οργανώσεις αλίας, την ΕΑΦ, την ΑΦΟ και την ΆΙΚΑΤ και σε κάποιες από αυτές σε συγκεκριμένα είδη. Στην ΆΙΚΑΤ, για παράδειγμα, επικεντρώνεστε μόνο στον ερυθρό Εγώ θα ήθελα να ξέρω και επιπλέον η σχέση με τρίτες χώρες είναι και σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινείται η υπηρεσία ελέγχου. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον στο μέλλον θα μπορούσαμε να διαβρεθούμε και σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις αλίας ε, στις οποίες ε, διαπιστώνονται προβλήματα και από ό,τι καταλαβαίνω ε, με κάποιες από αυτές είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα της λαθρέας και παράνομης αλίας και θα μπορούσατε λοιπόν να εκταθείτε και σε άλλα είδη για τον ερυθρό τόνο γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα αλλά υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται και σε, για άλλα είδη που έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από τον ερυθρό τόνο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν κατά πόσον θα γίνουν λίγο πιο ευέλικτα τα πράγματα στο μέλλον και θα διευρυνθούμε και σε άλλες περιοχές σε άλλους τομείς και σε άλλες τρίτες χώρες. Και επίση, με βάση αυτά που ρώτησε και ο κύριο Σάντσε Πρεσέδο, έχω και εγώ μια ερώτηση. Στην μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική υπάρχει ε, θέμα επέκτασης ε, της έρευνας ε, σε θέματα λίας. Μπορείτε εσείς να επεκταθείτε και σε θέματα αυτά υπάρχει κάποια υπηρεσία που μπορεί να συντονίσει την αλληλευτική έρευνα που γίνεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι εσείς θα μπορούσατε ίσως να αναλάβετε αυτά τα καθήκοντα, ίσως με περισσότερο προσωπικό και κάποιο περισσότερο ε, πόρους στη διάθεσή σας, αλλά επειδή ακριβώς συζητάμε τα θέματα της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να βρούμε και κάποιον ο οποίος θα συντονίσει τα θέματα της ε, αλληλευτικής έρευνας και θεωρώ ότι η υπηρεσία σας είναι πλέον ενδεδειγμένη για να ε, υλοποιήσει αυτή τη, αυτό το καθήκον. Έχετε το λόγο όμως, θα μας πείτε και εσείς περισσότερο. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω με τη δική σας ερώτηση για το θέμα της έρευνας. Ε, δεν προβλέπεται αυτό από τον κανονισμό ίδρυσης της υπηρεσίας. Βεβαίως είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ερώτημά σας, κυρίως διότι γνωρίζετε πως υπάρχει σοβαρή γύρανση των ερευνητών στον αλλιευτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα διατηρηθεί η τεχνογνωσία και πώς θα γίνει η ανταλλαγή ε, των γνώσεων, των στοιχείων που έχουμε σε σχέση με τα διάφορα αποθέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, γιατί επί τη βάση αυτών των στοιχείων λαμβάνονται και πολιτικές αποφάσεις. Ε, σήμερα ε, δεν μπορώ να σας απαντήσω καταφατικά, διότι σας είπα δεν προβλέπεται ε, στον κανονισμό ίδρυσης της ε, υπηρεσίας, ε, ούτε και στον εσωτερικό μας κανονισμό και σίγουρα χρειάζονται σημαντικά κονδύλια και ανθρώπινη πόροι για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Αλλά πάντως, ε, αν αλλάξει η κατάσταση, θα βελτιωθεί η κατάσταση ως προς τη διαμόρφωση επιστημονικών απόψεων ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόθεση αυτών στα διεθνή φόρα. Για τις σχέσεις με τις υπόλοιπες ζώνες, είναι προφανές ότι η υπηρεσία εργάζεται επί τη βάση ενός πρώτερου προγράμματος επιθεωρήσεων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είναι σαφές ότι ως προς την περιφερειακή διάσταση θα καλύψουμε και άλλα είδη. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά ε, θέλουμε να καλύψουμε την συντριπτική πλειοψηφία ε, των ειδών σε κάθε ζώνη, ούτως ώστε να μην ελέγχουμε μόνο ένα απόθεμα, αλλά να ε, προσεγγίζουμε το θέμα σφαιρικά, διότι πρόκειται για οικονομίες κλίμακας, και ε, θα πρέπει να αποτρέψουν αυτές τις ε, παρατυπίες ε, που εμποδίζουν την υλοποίηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η κυρία Λόνες από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ κρίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και κυρίως το θέμα της διαθεσμικής ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με όλα τα θεσμικά όργανα που είναι συναρμόδια, ΕΜΣΑ, Frontex, Παραδείγματο χάρη, Επίσης, συνεργασία με την υπηρεσία της Ιρλανδίας για τα κτηνιατρικά ζητήματα μπορεί να μας βοηθήσει πολύ ως προς τους ελέγχους DNA που ανέφερε η κυρία Λαβίν. Υπάρχουν δυνατότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες ε, κυρίως εντοπίζεται στη λεκάνη Μεσογείου ε, με τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, με την Τουρκία, τη Ρωσία στα, για τη Βαλτική και φυσικά με τον Καναδά. είναι υπαρκτές ε, αυτές είναι δυνατότητες, όμως θα πρέπει να εγγραφούν σε ένα ε, αρκετά επίσημο θεσμικό πλαίσιο. Για τις διεθνείς σχέσεις και τους πόρους, τα μέσα που διαθέτουμε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στην κυρία Λεβίν. Το θέμα του σκάφους που ε, ναυλώσαμε είναι, ξέρετε, και συμβολικό το θέμα. Πρόκειται για τη διεθνή διάσταση, αν θέλετε, της κοινής ελευθερικής πολιτικής. Ε, συμβολίζει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπροσωπείται ικανοποιητικά ε, στις εξωτερικές σχέσεις. Τώρα, ε, ως προς επιθεωρήσεις εν πλώ και ε, κατά την εκφόρτωση, δεν ελέγχουμε τα ίδια πράγματα. Η θαλάσσια επιθεώρηση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας επιτρέπει να εντοπίζουμε παρατυπίες ως προς τα τεχνικά μέτρα Επίσης μας επιτρέπει να ελέγχουμε σε πραγματικό χρόνο ε, τους ε, κανόνες που διέπουν ε, τα αλλιεύματα, κυρίως ως προς το μέγεθος των ματιών των δικτυών που είναι μεγαλύτερο που προβλέπεται στη συγκεκριμένη ζώνη. Τώρα κατά την εκφόρτωση κάνουμε άλλου είδους ελέγχους. Ελέγχουμε το βάρος, την ποσότητα και ε, διαπιστώνουμε κατά πόσο είναι ειλικρινείς ε, οι δηλώσεις γιατί έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικά εργαλεία ε, στην διάθεσή μας. Είναι δύο πυλώνες που συνυπάρχουν, η έλεγχη εν πλώ και η έλεγχη κατά την εκφόρτωση. Για την εκφόρτωση, όταν τροποποιήθηκαν τα συστήματα ελέγχου, επιφέραμε αλλαγή, γιατί δεν πρέπει να ελέγχουμε τις ποσότητες που εκφορτώνεται, φυσικά είναι σημαντικό, αλλά και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι θα αντικαταστήσουμε τους ελέγχους εν πλώ, γιατί για ήδη όπως ο ερυθρός τόνος είναι ε, απαραίτητη αυτή η έλεγχη. Για την Μεσόγειο, ζητώ συγγνώμη, μάλλον δεν ήμουν σαφής για αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντική η Μεσόγειος για την υπηρεσία μας, κυρίως για τον ερυθρό τόνο και η ΆΙΚΑΤΕ επικύρωσε και μία σύσταση για τον Ξηφία πρότεινε να ενταχθεί στο κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον ερυθρό τόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Μεσόγειος είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η διεπαφή αν θέλετε ανάμεσα στο βορρά και στο νότο και η σχέση και ε, ε, ο σύνδεσμός μας ενώνει με την ICAT και άλλες περιφερειακές οργανώσεις. Επίσης, ε, είναι, ο σύνδεσμός μας κατοχυρώνεται έτσι σχέση μας με όλες τις παράκτιες της Μεσογείου χώρες, είτε είναι στο βορρά είτε στο νότο της Μεσογείου. On se base part ε, ε, τώρα, θα ήθελα να ε, σχολιάσω λίγο το θέμα των ελέγχων. Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση κινδύνου, αλλά είναι αδύνατον να ελεγχθεί ένας οικονομικός τομέας αν δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, η βιομηχανία πρέπει να ξέρει με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί ο έλεγχος για να γίνει δεκτός από τους ελεγχόμενους οι επαγγελματίες πρέπει να ε, κατανοήσουν τις τεχνικές ε, λεπτομέρειες ε, του ελέγχου, αλλά πρέπει να θεωρήσουν επίσης ότι ο έλεγχος τους προστατεύει ενάντια των ανταγωνιστών που δρούν με αθέμητους όρους. Στο 90% των περιπτώσεων δεν είναι σίωση έλεγχοι, δεν υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς σε εισαγωγικά. Βεβαίως, όπως είναι αναμενόμενο για τους ελέγχους, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό άρνησης, παραδείγματος χάρη των ελέγχων ή επιθετική συμπεριφοράς Ε, εμείς έχουμε και μια συμβουλευτική υπηρεσία ε, για τις σχέσεις ε, με τον κλάδο και τις σχέσεις με τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Εφόσον μιλάμε για, την αρμοδιότητα εθνική ως προς τις άδειες, θα προσέθετα μόνο ότι ε, ε, προσπαθούμε να ε, εφαρμόσουμε ομοιόμορφους όρους ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, θέλουμε με τις δράσεις μας να κατοχυρώνουμε ισότιμη μεταχείριση για όλους αλληλείς. Θέμα τώρα παρακολούθησης των σκαφών. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει για την υπηρεσία μας. Και τώρα θα επανέλθω γενικότερα στο θέμα των, μέσων, των ελεκτικών μέσων που διαθέτουμε και του ναυλωμένου αυτού σκάφους. Μέσω της κρίσης είναι δύσκολο να ζητήσουμε περισσότερα πράγματα από τα κράτη-μέλη. Ε, η εξαφάνιση αυτού του ε, σκάφους ε, το 2012 θα αντικατασταθεί από κάποιες ε, αυξημένες εθνικές προσπάθειες, κάποια περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβόλαια και αυτό προκύπτει από το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ελέγχου σε σχέση με τα αλληλευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του κράτους. Στα πλαίσια της ICAT σε λίγες εβδομάδες μήνες θα προταθεί αυτό το σύστημα. Στην ΕΑΦΚ ήδη σημαίνει. Ε, όμως πρέπει να συνυπολογίσουμε το κόστος του ελέγχου να διαθέτουμε συστήματα παρακολούθησης μέσω δορυφόρου, διάδοσης ε, πληροφοριών, να διαθέτουμε συστήματα που μας επιτρέπουν να ε, γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο ή ελαφρώς διαφοροποιημένο χρόνο το τι κάνει το κάθε σκάφος, στοιχεία ε, επιστημονικά, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το κόστος ε, των ελέγχων σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Δεν θα ήθελα να ξεχάσω τώρα που δίνω τις απαντήσεις μου το ζήτημα της ε, παρουσίας των ε, νοσιακών σκαφών στα λιβικά είδατε. Δεν ξέρετε ότι η Λιβύη έχει ε, την εξή ιδιαιτερότητα ότι στον κόλπο της Σύρτης ε, δεν είναι ξεκαθαρισμένα τα ε, διεθνή ύδατα, το εύρος των διεθνών υδάτων και έχουμε και την συνθήκη της Βενετίας του 83 που έχει προβλέψεις για τη συγκεκριμένη ζώνη. Κάποια κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν αυτή τη σύμβαση ε, και θεωρούν ότι εκεί στον κόλπο της Ήρτης είναι διεθνή τα ύδατα. Αυτό ισχυρίζονται και αλλιεύουν εκεί. Υπάρχουν σκάφη με σημαία της Λιβύης, αλλά ε, που ναυλώνουν ε, οι υπήκοοι της Ένωσης και άρα διαφεύγουν, εκφεύγουν από αυτά τα μέτρα διατήρησης των αποθεμάτων, αλλά αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Ε, και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη δράση του επόπτη προστασία ε, των ε, προσωπικών δεδομένων. δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε δηλαδή κάποια στοιχεία. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε κύριε Ρομέντα αλλά στον τομέα αυτό τη εφαρμογή κοινή αλληλευτική πολιτική, νομίζω τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν πιο σημαντικέ προσπάθειες. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα στον πιθανό ελεγκτικό ρόλο της υπηρεσίας ως προς τα κράτη-μέλη. Σας παραπέμπω στη συνθήκη. Ο θεματοφύλακας των συνθήκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρει και την ευθύνη για την εφαρμογή της κοινής ελευθερικής πολιτικής, έχει ε, την ευθύνη ελέγχου των ε, κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των ε, ε, διαδικασιών επί παραβάση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ένωσης. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, η υπηρεσία είχε ως στόχο την ενίσχυση του συντονισμού της συνεργασίας. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να είμαστε και δικαστές και κατηγορούμενοι, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε το συντονισμό και ταυτόχρονα να ελέγχουμε και τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται διεύρυνση εν αυτή η περιπτώση της αρμοδιότητας της υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε πόσο λεπτό είναι αυτό το ζήτημα και υπερβαίνει κατά πολύ τη θέση μου, την αρμοδιότητά μου. Τέλο πάντων, ε, για να κλείσω αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ε, στην αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κανονισμός 1224 ε, του 2009 για την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ε, προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις για τους εμπλόκοι και επίγειους ελέγχους. Οι επίγειοι ελέγχοι έχουν ε, σημαντική έχουν σημαντικό ρόλο ως προς την περαιτέρω ε, θέση σε εμπορία των προϊόντων και ως προς την ε, ανιχνεσιμότητα των προϊόντων γιατί αυτό είναι σημαντική συνιστόση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Σήμερα οι επίγειοι έλεγχοι που εντάσσονται στα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα περιορίζονται στη φάση εκφόρτωσης. Ορισμένες φορές μπορούμε να ελέγξουμε τα προϊόντα κατά τη μεταφορά, αλλά ε, ούτως ή άλλως ε, το σχέδιο της επιθεώρησης ε, και του ειδικού αυτού ελέγχου προβλέπει τον τόπο ελέγχου αν θέλετε. Στα προγράμματα εργασίας των κρατών μελών υπάρχουν κάποια σχετικά στοιχεία και το ταχύτερο δυνατόν θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα επίσης. Στη CGP PM και στην ΆΕΚΑΤ έχουμε κάνει σχετικές συνεδριάσεις. Στις αρχές του 2012 έχουμε μία συνεδρίαση CGPM για τον εύξηνο πόντο όλα τα παράκτια ε, κράτη θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συνεδρία του Ιανουαρίου. Τώρα για την ε, μελλοντική αλληλευτική πολιτική είμαστε στη διάθεση του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και με, υπό την επιφύλαξη των μέσων που έχουμε θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και ως προς τα τεχνικά μέτρα για την απαγορεύση των απορρίψεων, παραδείγματος χάρη ή οποιαδήποτε άλλα ε, μέτρα αποφασιστούν βάσει αυτή τη νομοθετική διαδικασία, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όλα αυτά τα νέα τεχνικά μέτρα θα σα βοηθήσουμε να τα εφαρμόσετε. Και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τόσο αναλυτικές ε, πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ ε, εκ νέου για την παρουσία σας εδώ. Επιβεβαιώνω ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία που θα επισκεφθεί την υπηρεσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστή και ο Bueno, con esto el señor Romeva desaparecido. Ο κύριο Ρωμέβα εξαφανίστηκε. Όχι, νάτος. Ελάτε, ελάτε να μα τα πείτε για τον ερυθρό τόνο. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη και περνάμε στο σημείο υπαριθμών 8. Τροποποίηση του κανονισμού υπαριθμών 302-2009 για τη θέσπιση πολιετίου σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, σχέδιο αποκατάστασης που εγκρίθηκε πέρσι στο Παρίσι το συζητάμε σήμερα και όχι πριν από κάποιες εβδομάδες, ε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η νέα συνεδρίαση της ICAT στην Κωνσταντινούπολη και υπήρχε περίπτωση να υπάρξουν τροποποίησεις. Δεν έγιναν τροποποίησεις επί της ουσίας, αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να λάβουμε υπόψη και αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό λοιπόν παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε τροποποιήσει επί τη ουσία, υπήρχαν κάποιες αποφάσεις τεχνικού χαρακτήρα, τις οποίες θεωρώ και θετικέ σε κάποιες περιπτώσεις. Όσον αφορά τη μεταφορά που πρέπει να κάνουμε εμείς ε, στο κοινοτικό κεκτημένο, δεν ε, ήταν ιδιαίτερα ουσιαστικέ οι αλλαγέ. Η πρότασή μου τώρα έχει σχέση καταρχάς με την ανάλυση της κατάστασης και κατά δεύτερον με τα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε ε, σε αυτή τη συμφωνία. Η ανάλυση της κατάστασης να εξηγήσω δύο-τρία πράγματα και καταρχάς δεν θα πρέπει να λύσμονουμε ότι η κατάσταση του ερυθρού τόνου είναι πολύ ευαίσθητη Πρόκειται επίσης και για το είδος το οποίο φυσικά έχει περισσότερες δυνατότητες ε, ρύθμισης, ε, αν όχι σε παγκόσμια κλίματα, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δούμε την νομοθεσία και τα μέτρα τα οποία ρυθμίζουν ε, την διαχείριση του ερυθρού τόνου και τα συγκρίνουμε με είδη τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και σε κάποιες περιπτώσεις ε, ε, ακόμα χειρότερη, είναι ουσιαστικά τα μέτρα. Πρόκειται για ένα είδος αλληλείας το οποίο είναι πάρα πολύ ρυθμισμένο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επαρκούν τα μέτρα αυτά για τους στόχους που προσπαθούμε να επιτύχουμε κυρίως διότι εξακολουθούμε να έχουμε διαθροτικά προβλήματα, να υπάρχει υπεραλίευση, να υπάρχει έλλειψη ελέγχου, να υπάρχει παράνομη αλία, να υπάρχει κακή πληροφόρηση ή λανθασμένη πληροφόρηση, με, να υπάρχουν προβλήματα τα οποία πολλές φορές σχετίζονται στην, με την μη τήρηση της νομοθεσίας και ούτω καθεξής. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πριν από ένα-δύο χρόνια υπήρξε μια ανεξάρτητη έκθεση η οποία αξιολόγησε κατά την άποψή μου ε, κατέδειξε και ιδιαίτερα ανησυχά, ανησυχητικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η ICAT τον ερυθρό τόνο και είπε ότι είναι ε, παγκόσμιο όνειδος ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει, διότι η υπερβολική νομοθεσία δεν σημαίνει απαρατήτως ότι γίνονται όλα σωστά σε αρκετές περιπτώσεις. Είδαμε σήμερα κάποια στοιχεία για το ε, έτος που μας πέρασε, για τους ελέγχους που διεξήγαγε η υπηρεσία. Κάποια από τα στοιχεία ε, μας έδειξαν ότι είχαμε κάποιες περισσότερες ε, ε, ελεγκτικές διαδικασίες από το 2010 που είχαμε μόνο 7 ελέγχους, είχαμε περισσότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιλύσαμε το πρόβλημα. Βελτιωθήκαμε μεν, αλλά πόρα απέχουμε από την επίλυση των προβλημάτων. Αυτός προς την ανάλυση. Τώρα, αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή είναι η εφαρμογή των όσων εγκρίθηκαν από πλευρά ICAT και αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Όπως για παράδειγμα το γεγονός της μείωσης των τάκ και των ποσοστώσεων ιδίω τον ΤΑΚ, ε, το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα, ως προς τις ποσότητες που εκτιμάται ότι μπορούμε να αλλιεύσουμε νομίμως και Υπάρχει, υπάρχει και μια μικρή συζήτηση εδώ για το κατά πόσον επαρκεί αυτή η ποσότητα, αυτό το ΤΑΤ για να επιτευχθούν ε, οι στόχοι της αποκατάστασης του είδου. Ε, αυτή βέβαια είναι επιστημονική συζήτηση. Ε, κάποιοι εξημών που είμαστε πιο συντηρητικοί ε, θεωρούν ότι επαρκεί, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν είναι επαρκές. Αλλά το θέμα είναι ότι το ΤΑΤ έχει εγκριθεί και πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι πιο τεχνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα πώς ε, γίνεται ο έλεγχος, ε, η παρουσία των ε, επιθεωρητών και παρατηρητών επί των σκαφών και σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς αλλιευτικών για κάποια θυναλιευτικά και τράτες. Θα πρέπει επίσης να θέσουμε και το θέμα ουσίας. Το κατά πόσον αυτό το σχέδιο αποκατάστασης θα μας επιτρέψει να έχουμε ανασύσταση του είδους που είναι αυτό που επιθυμούμε. Το πρώτο θέμα, και γι' αυτό και προτείνω και σχετική τροπολογία, κατά πόσον μπορούμε να θέσουμε αποκατάσταση βάσει του BMSY ε, της βιομάζας ε, δηλαδή στο μέγιστη βιώσιμη απόδοση στο σχέδιο αποκατάστασης προβλέπεται να έχουμε 60% αποκατάσταση του BMSY μέχρι το 2022. Αυτό είναι μέσω της ICAT που είναι διεθνές πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένες νομοθεσίες ε, για παράδειγμα στην οδηγία για την θαλάσσια στρατηγική ε, υποχρεούμεθα να έχουμε ένα καλό περιβαλλοντικό επίπεδο, δηλαδή ένα καλό BMSY για το 2020. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και δεν συμπίπτει απαραίτητο με αυτό το οποίο εγκρίθηκε σε διεθνές επίπεδο. Και επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένε δεσμεύσεις με τη δήλωση του Johannesburg, στην οποία καθορίζεται ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι ε, να επιτύχουμε το BMSY το 2015. Ε, Και ε, λέμε μεν ότι δεν έχει σχέση από πολιτική σκοπιά, εγώ όμως κάνω τη διάκριση και λέω ότι άλλο είναι το διεθνές πλαίσιο και άλλο είναι οι διεθνής δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τηρούμε τα όσα έχουμε υπογράψει όταν πηγαίνουμε σε άλλες διεθνείς ε, επισκέψεις. Η πρώτη λοιπόν εκ των τροπολογιών που κατέθεσα και θεωρώ ότι συνάδει με τη μεταφορά της νομοθεσίας της ICAT είναι μια τροποποίηση για το επίπεδο ε, πιθανοτήτων ε, και την επίτευξη του BMSY. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τονίσω εδώ, είναι ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στην ICAT κατά την άποψή μου δεν είναι άσχημα αλλά είναι ανεπαρκή. Δεν είμαι αντίθετος ε, στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, απλώς θεωρώ ότι απέχουν απέχουν μακράν των όσων προσπαθούμε να επιτύχουμε. Είναι απαραίτητα, ανεπαρκή μεν αλλά απαραίτητα. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει και μπορούμε να τα υιοθετήσουμε λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός αυτό, ότι πρέπει να τα συμπληρώσουμε και με άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο φιλόδοξα σε κάποιες συγκεκριμένε περιοχές. Και εγώ προτείνω δύο μέτρα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι εφικτά και ε, είναι και κατεπήγοντα, όχι μόνο απαραίτητα. Το πρώτο να έχουμε τις λεγόμενες περιοχές οτοκίας. Περιοχές ε, στις οποίες θα υπάρχει προστασία και κατά βάση θα διασφαλίζεται ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει οτοκία και αναπαραγωγή του ερυθρού τόνου και δηλαδή ε, ε, δίνεται προστασία ώστε να διασφαλίζεται αυτή η δραστηριότητα. Ο χάρτης είναι καθορισμένος, είναι σαφής και το σχέδιο που έχω είναι ε, η τροπολογία μου δηλαδή είναι να έχουμε αυτές τις έξι περιοχές οι οποίες θεωρούνται ευαίσθητες περιοχές και αναφέρομαι κυρίως στις ε, ευρωπαϊκές ε, περιοχές από περιφερειακή σκοπιά αλλά και για τα σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία που δραστηριοποιούνται εκτός ευρωπαϊκών υδάτων. Το δεύτερο μέτρο που προτείνω είναι η άρση μιας παρέκκλησης για την Αδριατική θάλασσα, η οποία επιτρέπει να αλλιεύονται τόνοι 8 κιλών ενώ η οδηγία απαιτεί 30 ε, κιλά διότι κατά βάση αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η παρέκκληση αυτή ε, χρησιμοποιείται από τα βιομηχανικά σκάφη και ορισμένες φορές είναι λανθασμένη η χρήση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σταματήσει να ισχύει η παρέκκληση. Πρόκειται για δύο μέτρα τα οποία είναι πολύ απλά και πολύ εύκολο να υλοποιηθούν, γι' αυτό ακριβώς και τα προτείνω. Ως ε, εισηγητής ε, θα πρέπει επίσης να τονίσω αυτά τα οποία μας πρότειναν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, κυρίως την ε, συνάδελφο Τάβια Σάρτου. Υπάρχουν μια σειρά από συστάσεις τις οποίες εμείς ως Επιτροπή Αλίας θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και ε, κάποια σχετίζονται και με κάποια από τα πράγματα τα οποία προτείνω εγώ και επομένω ε, θα πρέπει να ε, τα προσθέσουμε γιατί σε κάποια στοιχεία πηγαίνουν και λίγο παραπέρα. Ε, θα είναι σίγουρα θετική η σύστασή μου σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως σε δύο στοιχεία. Πρώτον, η ανάγκη να ελέγχουμε καλύτερα ε, και ε, περισσότερο τα ηχθειοτροφία. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα το έχουμε κυρίως τα ηχθειοτροφία. Όχι μόνο ε, λόγω του υπολογισμού αλλά και του ελέγχου των ποσοτήτων που έχουμε στα ηχθειοτροφία. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από την ICAT που είναι η έγκριση του ηλεκτρονικού BCD. Καλά όλα αυτά, αλλά αυτό βελτιώνει μόνο τις ε, οδηγίες τις οποίες διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, τις πληροφορίες που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή και αντί να τις έχουμε σε χαρτί θα τις έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή. Το πρόβλημά μα όμως είναι τα δεδομένα. Δεν είναι το αν θα τα διαθέτουμε σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικό πλαίσιο. Θέλουμε να ξέρουμε ότι τα δεδομένα αυτά ανταποκρίνονται στα στοιχεία που πραγματικά έχουμε για τα εκθετορφία. Και εκείνο που είναι σημαντικό επίσης είναι να λάβουμε υπόψη ότι στον τομέα υπάρχουν τελείως διαφορετικές ευαισθησίες. Όταν αναφερόμαστε στον κλάδο, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις σε κάποιους συγκεκριμένου τομείς του κλάδου και αυτές οι τομείς οι οποίοι είναι πιο επιζήμοι και που έχουν πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις ε, για την αλληλεία θα πρέπει να ελέγχονται ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, ε, πολύ περισσότερο και να υπάρχουν πολύ περισσότερες κυρώσεις από ό,τι έχουμε σήμερα. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση βέβαια. Δεν έχω και κάποια πολύ νέα στοιχεία να διαβιβάσω από τα όσα έχουμε από την ICAT. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πιο διεξοδική ανάλυση και μπορεί να με διορθώσει. η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται και με τα σημαντικά στοιχεία που έχουμε από τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Υπάρχει και το θέμα του EBCD και πέρα από αυτά δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, εάν βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη, είμαι ε, όλος αυτιά για να το ακούσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει κάποιο το λόγο. Θα μιλήσω εγώ. Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεσή σας και πρέπει να σας πω καταρχάς ότι διαφωνώ με την τροποποίηση του σχεδίου πολιετούς ανασύστασης του ερυθρού τόνου μονομερός για τον ευρωπαϊκό στόλο. Συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής στη συνεδρίαση την ΆΙΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα ότι το πρόγραμμα αποκαταστασής ε, μένει ως όχι μέχρι νεοτέρας. Αυτό κατά την άποψή μου είναι η πιο ευφυής απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης διαφωνώ και με τις τρεις τροπολογίες που καταθέσετε και θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι η μονομερής τροποποίηση προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε ουσιαστικά καταδικάζει όλο τον κοινοτικό στόλο που αλλιεύει ερυθρό τόνο στη Μεσόγειο. Με φοβίζει όμως το γεγονός ότι θέτετε εσείς ένα 20% όταν η ΆΙΚΑΤ κατέλαβε απόφαση για το πολιετές ε, σχέδιο και η πλειονότητα των σχεδίων αποκατάστασης της ICAT έχουν 50% πιθανότητες με αποθέματα τα οποία ε, βρίσκονται σε πολύ πιο χειρότερη κατάσταση από τον ερυθρό τόνο. Να αποφασίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε διπλή επίθεση για τον ερυθρό τόνο δεν καταλαβαίνω προς τι μας εξυπηρετεί εάν δεχτούμε το 90% πιθανότητες που προτείνετε εσείς, θα σήμαινε ότι θα πρέπει να σταματήσει να ψαρεύει ο στόλος. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές ε, οτοκίας, εγώ ε, ασχολούμαι με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ε, σύσταση, η οποία να λέει ότι πρέπει αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές να είναι περιοχές οτοκίας, δεν ε, ε, διαπίστωσα και επομένω δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι. Όσον αφορά την τελευταία σα τροπολογία για τα ελάχιστα μεγέθη, θα μπορούσα να δεχτώ κάποια από τα επιχειρηματά σα, αλλά ε, επειδή η λογική μου είναι ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει τίποτα στο σχέδιο αποκατάσταση μέχρι νεωτέρας διαφωνώ λοιπόν και με αυτήν. Υπάρχει και η εξή αλλαγή. Φέτος στην ICAD εγκρίθηκε μια νέα επιστημονική ανάλυση για να δούμε πού βρίσκονται τα ε, αποθέματα του ερυθρού τόνου και θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε αυτή την επιστημονική γνωμοδότηση ε, πριν ε, λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση, ακόμα και αν πρέπει να πάμε στην κατεύθυνση που υποδεικνύετε εσείς. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε την ανάλυση λοιπόν για να λάβουμε μέτρα. Κύριε Ρωμέβα Ιρουέδα, λυπάμαι που διαφωνώ μαζί σας. Αυτή είναι η θέση μου. Να... Θα σας δώσουμε το λόγο. Ε, ο κύριος Ντονατέλα όμως έχει ζητήσει το λόγο καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα συνεχίσουμε. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να διευκρινίσω ορισμένε τεχνικές λεπτομέρειες. Ε, είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση αυτή με τα τεχνικά επιχειρήματα λόγω της πρότασης που έχουμε και πιστεύω ότι υπάρχουν εδώ πάρα πολλές λεπτομέρειες και δι τεχνικής φύσης. Επίσης, την τελευταία εβδομάδα η συνεδρίαση της ΕΚΑ 2011 ολοκληρώθηκε και συζητήθηκε ο ερθρός τόνος σε μεγάλο βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ μία σαφέστατη και βιώσιμη ε, πολιτική και αρνήθηκε να την τροποποιήσει είτε σε τυπική είτε σε ουσιαστική είτε στις τυπικές είτε στις ουσιαστικές πτυχές. Όσον αφορά τώρα την πολιτική πτυχή η Κομισιόν είπε ότι σε αυτόν τον τομέα αλλά και για τα όργανα ελέγχου είναι πολύ σημαντικό να εγγυηθούμε μια σταθερότητα στην ε, μεταρρύθμιση και δει στην εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης. Αυτό το λέει και ο εισηγητής στην έκθεση του και αυτό οδηγεί σε μια σταθεροποίηση έναντι και εκείνων που πρέπει να εξασφαλίσουν το εισόδομα τους αλλά και τη σωστή διαδικασία διενέργειας της αλίας. Όπως ακούσαμε και από την η ε, ε, υπηρεσία του Βίγκο είναι, στο Βίγκο είναι πολύ σημαντικό να διανεργούνται σωστά οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις. Το 2011-2012 θα υπάρχει μια πλήρης ε, ε, η εφαρμογή ενός απόλυτου σεβασμού της, ε, ε, του κανονισμού που θα εφαρμόζεται από τις διοικήσεις των κρατών μελών. Πρέπει να γίνει απόλυτα, απόλυτα σεβαστές οι διατάξεις του κανονισμού. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις ζώνες ανασύστασης και τον καθορισμό αυτών των ζωνών και των ζωνών αποκλεισμού αλίας, εδώ συντονίζουμε τις ε, προτάσεις μας ε, μαζί με την υπηρεσία του κυρίου Σαβουρέ, όπως είπε και ο ίδιος, και έτσι μπορούμε να παρέμβουμε σε ορισμένε διεθνείς περιοχές, διεθνείς ζώνες και εκεί μπορούμε να διενεργούμε όχι μόνο ελέγχους αλλά στοχευμένες ε, ενέργειες πάνω σε σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία αλλά και να παρακολουθούμε άλλες διατάξεις της ΕΚΑΤ. Το 2011 διενεργήσαμε περίπου 20 επιθεωρήσεις και διαπιστώσαμε ε, διενεργήσαμε 12 ελέγχους και διαπιστώσαμε 20 σοβαρές παραβιάσεις. Και το γεγονός ότι μπορούμε να ενεργούμε σε ζώνες οι οποίες με την αυστηρή ερμηνεία ας πούμε δεν εμπίπτουν στις ζώνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και μια ε, δυνατότητα πολύ σημαντική. Ε, και πρέπει να τη διατηρήσουμε διότι εάν εμείς πρέπει να υιοθετήσουμε μονόπλευρα μέτρα θα μπορέσουν ενδεχομένως ε, εφαρμόζοντας ε, αυστηρά την τυπική, τις τυπικές διατάξεις της να απαγορεύσουν την, την παρουσία μας σε αυτές τις αμφιλεγόμενες ζώνες ενώ εμείς θέλουμε να μπορούμε υπό το πλαίσιο της ΆΙΚΑΤ να διενεργούμε αυτές τις ε, ενέργειες ελέγχου, επισόρησης και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη σε κάθε συζήτηση που γίνεται διότι ε, ο στόχος μας είναι να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι ευαίσθητες ε, ζώνες αποκατάστασης και να μπορούν να διενεργούνται εκεί οι κατάλληλοι έλεγχοι. Ε, ε, αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ζώνες, σε περιοχές οι οποίες δεν εμπίπτουν αυστηρά ε, στην ε, δικαιοδοσία μας. Η ICAT μας έχει ζητήσει πολλές φορές τα συμβαλόμενα μέρη να εκτελούν τις, τους επιτρεπόμενους ελέγχους και να επισημαίνουν ε, και να ταυτοποιούν τις τυχόν παραβιάσεις ή παρατυπίες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η παρουσία μας σε αυτές τις ζώνες ε, ανασύστασης. Ο, εξετάζοντας τις προτάσεις ε, του εισηγητού, έχουμε να χειριστούμε θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κοινοτική νομοθεσία και βεβαίως υπάρχουν και επιχειρήματα τα οποία ε, είναι κατανοητά. Όμως υπάρχουν ε, και λεγόμενες γκρίζες ε, ζώνες, αφιλεγόμενες και αμφισβητούμενες περιοχές ή ζητήματα. Υπάρχουν ζώνες στην περιοχή της Μεσογείου όπου αμφισβητείται ακριβώς που εμπίπτουν και πώς ερμηνεύεται και ε, πώς ερμηνεύονται διατάξεις ε, πάνω σε, σε, αυτές τις περιοχές. Ε, υπάρχουν και θέματα εθνικής κυριαρχίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την πρόσβαση σε αυτές τις ζώνες, έστω και αν είναι αφυλακόμενες, διότι οι εταίροι μας το, το το επισημούν αυτό πολύ, το ε, ιδιαίτερος. Και γι' αυτό essentiel en tout cas pour la Commission, c'est la nécessité d'assurer dans le futur une... Euh, Και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη στο μέλλον να διατηρηθεί αυτό το πρόγραμμα ελέγχου, ειδικά επειδή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στα αξιοτροφία. Η κυρία Δαμανάκη το είπε αυτό, ότι οι έλεγχοι στις περιοχές των ιχθυοτροφίων θα αποτελέσουν ένα κεντρικό σημείο του προγράμματος του 2012. Και γι' αυτό επίσης θέλουμε οπωσδήποτε να ενισχύσουμε και να εξασφαλίσουμε το συνολικό πρόγραμμα ελέγχων. Αυτό εγγράφεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι έχει προβλεφθεί ήδη ενίσχυση ε, αυτού του στοιχείου ελέγχου στο τωρινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριο Ρουέντα. Ναι, για να διευκρινίσω ένα-δυο πράγματα. το να λαμβάνουμε μονομερείς αποφάσεις, από ό,τι ξέρω είναι περίπλοκο, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε και ένα ουσιαστικό στοιχείο, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για το 56% του τάκ του ερυθρού τόνου. Ουσιαστικά λοιπόν έχει ηγετικό ρόλο να διαδραματίσει ενώπιον των υπολείμων συμβαλωμένων ε, μερών και κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι ίσονο σημασία. Πρόκειται για σημαντικό θέμα και νομίζω ότι δεν ισχύει το ότι αν το κάνουμε εμείς ε, θα βγούμε χαμένοι. Ε, είναι λάθος αντίληψη αυτή του κλάδου έχουμε ευθύνη για την αποκατάσταση των αποθεμάτων και μάλιστα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα συμβαλωμένα μέρη, ε, των οποίων από ποσοτική κοπιάς ε, η επιρροή είναι πολύ μικρότερη. Επαναλαμβάνω λοιπόν τη θέση μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τον ηγετικό ρόλο και στη συνεδριάση τη ICAT και στην εφαρμογή των όσων εγκρίνονται στην ICAT. Δεύτερον, όσον αφορά το ποσοστό, το ποσοστό της πιθανότητας σε σχέση με την αποκατάσταση. Το πρόβλημά μου, το αναγνωρίζω, είναι κυρίως ονειολογικό. Ξέρω ότι συνήθως οι πιθανότητες τίθεται σε ένα επίπεδο της τάξης του 50-60%. Το ερώτημα που τίθεται κατά την άποψή μου και ξεκινώ και από τη βάση, τη γενικότερη κατανόηση του ζητήματος, είναι κατά πόσον εμείς ως πολιτικοί διαχειριστές έχουμε την πολυτέλεια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να έχουμε τόσο χαμηλά ποσοστά αποκατάστασης, πιθανότητε αποκατάστασης. Δεν ξέρω αν κάποιο από εσά θα ανέβαινε σε ένα αεροπλάνο, αν του έλεγα ότι έχει 550 ε, συγγνώμη, 60% πιθανότητα να φτάσει στον προορισμό του. Κανένας δεν θα έπαιρνε αεροπλάνο σε αυτή την περίπτωση. Και εγκρίνουμε προγράμματα αποκατάστασης με τέτοιες πιθανότητες δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, δεν είναι γελίο και θα πρέπει να τοποθετηθούμε πάρα πολύ σοβαρά. Τι ποσοστά πιθανότητας είναι λογικά για να εγκρίνουμε κάποια σχέδια αποκατάστασης, γι' αυτό ακριβώς και κάνουμε εμείς την πρόταση να φτάσουμε τουλάχιστον στο 90%. Θεωρούμε ότι είναι θέμα ουσίας ε, για την εφαρμογή ενός ε, σχεδίου και είναι και ε, ενιολογικό. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τον ερυθρό τόνο. Σημειώνω και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας έλεγε ο κύριος Ντονατόλα για το γεγονός ότι η παρουσία ευρωπαϊκών σκαφών σε διεθνή ύδατα είναι ακριβώς επειδή υπάρχουν σκάφη που θέλουν να αλλιεύουν σε αυτές τις περιοχές. Εδώ να σας κάνω το αντίστροφο επιχείρημα. Η παρουσία αυτή χρειάζεται για να ελέγχει όλη την αλλιευτική δραστηριότητα σε επαρκή βαθμό ώστε να είναι αυτό που θέλουμε το αποτέλεσμα ή όχι. Διότι ε, αυτό που μου λέτε ως αιτιολόγηση το κατανοώ. Αυτό που δεν είναι σαφές για μένα όμως είναι κατά πόσον επειδή καταγγέλλονται και συγκεκριμένα ποσοστά υπεραλίευσης είναι τόσο λογική η παρουσία των ελέγχων που έχουμε. Και ολοκληρώνω με το εξής. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί τροφή για σκέψη. Η έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε προσπάτως... Ε, το γεγονός ότι το 2015 θα έχουμε ένα τάκ 13.500 τόνων αιτιολογεί το γεγονός ότι ε, υπήρξε εμπορία 32.000 τόνων. Δηλαδή, Αυτοί οι 32.000 τόνοι ε, που τίθεται σε εμπορία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλοι στο ίδιο χρονικό διάστημα. Κάποιες μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές, ε, περιόδους αλίας. Αλλά παρά το γεγονός αυτό υπάρχει μια λογική αμφιβολία την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το σημείο κίνησης και γι' αυτό κάποιοι εξημών είμαστε τόσο απαιτητικοί για την τήρηση της νομοθεσίας. Πέραν αυτού βέβαια η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Αν δεν κάνω λάθος η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή και επομένως το Δεκέμβριο θα υπάρξει και η επίσημη θέση της Επιτροπής Αλίας και νομίζω ότι τον Ιανουάριο μπορεί το θέμα να περάσει και από την Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτό το τελευταίο σημαντικό σημείο που υπενθύμησε ο κύριος Δρομέντα. Όντω υπάρχουν δυσκολίες σε σχέση ε, με την διασταύρωση ε, στοιχείων που προέρχονται από τα BCD και από τα στοιχεία λιευμάτων, αφενός ε, και αφετέρου τα στοιχεία από τη θέση σε εμπορία. Από τότε που πήραμε στοιχεία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις άμεσα, αμέσως ζητήσαμε λεπτομερή έρευνα, ήρθαμε σε επαφή με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αναλύσαμε τα δεδομένα που υπήρχαν στην ιστοσελίδα της ICAT. Υπάρχει μια έλλειψη συνοχής ε, ανάμεσα σε, αυτά, σε αυτές τις δύο δέσμες ε, στοιχείων και στην Κωνσταντινούπολη ε, κάναμε ε, πολλές συνεδριάσεις ε, με την ΕΠΙΟΥ για να δούμε ποια μεθοδολογία χρησιμοποιούσε ο οργάνος για να καταλήξει αυτά τα στοιχεία. Ε, η σημερινή κατάσταση δεν είναι σαφής, διότι ακόμη επεξεργαζόμαστε τη μεθοδολογία και εκκρεμούν διάφορα ζητήματα. Ε, στο μυαλό μας υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, δεν είναι άμεσα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα γιατί οποιαδήποτε μεθοδολογία και αν χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιούμε διαφορετικές πηγές και διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας των δεδομένων. Ε, παρακολουθούμε πάντως από κοντά αυτό το φάκελο και θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και τους δύο. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 28 Νοεμβρίου. 12 το μεσημέρι. Ωραία. Ολοκληρώθηκε και το σημείο υπαριθμών 8 και περνάμε στο σημείο 12. Πολιετές σχέδιο για το απόθεμα Σολομού της Βαλτικής και την αλλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος. Ο κύριος Γκρόμπαρτσικ ε, είναι εισηγητής. Έχετε το λόγο. η θελετε να μιλήσει πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων για την εδραίωση ενός πολιετού σχεδίου για τα αποθέματα Σολομού της Βαλτικής. Θέλω να κάνω μια γενική παρουσίαση του θέματος, αλλά καταρχάς θέλω να ακούσω τη δική σας γνώμη και τη δική σας προτάσεις για το τι θέλετε να συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση. Θα αρχίσω αναφερόμενο στην κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα. Πριν από δύο χρόνια ή τρία χρόνια Στη Βαλτική θάλασσα η κατάσταση ε, ήταν παρόμοια με την έρημο όσον, αφορά τον γάδο. Ε, ε, και όλοι το είχαν αναφέρει αυτό, την απερίμωση της Βαλτικής από το γάδο και μειώθηκαν σημαντικά τα τάκ και αυτή η αποψήλωση του πληθυσμού του γάδου ήταν πολύ ενισχυτική και μετά από δύο χρόνια το Συμβούλιο αύξησε τα επιτρεπόμενα αλλιεύματα δύο και τρεις φορές και δυστυχώς ε, δίνεται εικόνα ότι δεν είναι πλέον ο γάδος είδος ε, που κινδυνεύει όσον αφορά δε τις αρτέλες... Ε, θεωρούνται πλέον ε, ε, κατάλληλες μόνο για, για τα ηχθιοτροφία, τροφή δηλαδή άλλων ειδών και όχι ως σημαντικό είδος κατανάλωσης, ηχθιάλευρα, για τα ηχθιέλεα. Το Συμβούλιο λοιπόν με την πρόσφατη απόφαση του είπε ότι θα ε, πρέπει να μειωθούν τα, τα επόμενα λιεύματα και πάλι ε, σημαντικότατα. Η ίδια κατάσταση ισχύει και για το Σολομό. Πρόσφατα το Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τα ΤΑΚ ε, σημαντικά, δραματικά και τίθεται το ερώτημα τι επιτέλους συμβαίνει. Περί πρόκειται εδώ. Προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον προσπαθούμε να προβλέψουμε τον καιρό, τι θα γίνει στο μέλλον, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία να βασιστούμε. Διότι αυτό το πολιετές πρόγραμμα για τα αποθέματα του λωμού στη Βαλτική υπάρχει και πρέπει να επισημάνουμε, να ταυτοποιήσουμε ε, τα αίτια για την μείωση των αποθεμάτων σολομού. Η διαδικασία που προβλέπει η Κομισιόν να ξεκινήσει έχει ακριβώς αυτούς τους στόχους, αλλά οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν ξέρουμε τους λόγους μείωσης των επιθεμάτων. Ξέρουμε για το γάδο τι συμβαίνει, ε, ξέρουμε για τη σαρδέλα τι συμβαίνει, ε, ε, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι κινδυνοί, πολλά άλλα είδη που κινδυνεύουν και δεν ξέρουν, δεν έχουμε πολλά στοιχεία παρά οι αλλοί μας ε, δίνουν ορισμένες πληροφορίες, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι ε, βάσιμες ε, και αξιόπιστες. Αναφέρουμε βεβαίως τη μείωση των πληθυσμών. Ειδικά για το Σολομό πρέπει να ερευνήσουμε τους λόγους μείωσης των πληθυσμών, διότι αν θέλουμε την αποκατάσταση, ε, πρέπει να φροντίσουμε πρώτα τη διατήρηση του υπάρχοντος αποθέματος στη Βαλτική θάλασσα. Ε, πρώτα διατήρηση, μετά αποκατάσταση. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίες, ε, από τη μία πλευρά έχουμε τους αλείς που μας δίνουν τις πληροφορίες, απ' την άλλη έχουμε περιβαλλοντολόγους και άλλους αρμόδιους φορείς που μας δίνουν στοιχεία περιβαλλοντικά, τα οποία έχουν επίπτωση στον σολομό της Βαλτικής. Και ε, έχουμε και ορισμένες πληροφορίες που λένε ότι τα αποθέματα αυξάνονται. Δεν υπάρχει λοιπόν μία βάσιμη αξιολόγηση των κινδύνων. Οι αλλοί λένε ότι ο πληθυσμό της ε, φώκιας ε, στη Βαλτική είναι τεράστιος, αλλά σύμφωνα με επιστήμονες η φώκια είναι ακριβώς ο μεγαλύτερος κίνδυνος, είναι ο μεγαλύτερος κυνηγός του Σολομού οι φώκες λατρεύουν το Σολομό και αυτό το στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ε, ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις των φυσικών συνθήκων στα αποθέματα Σολομού εάν ε, συμβαίνει πράγματι ότι οι φώκες είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ή ότι ο πληθυσμός της φώκιας επηρεάζει τον πληθυσμό του Σολομού, πρέπει οπωσδήποτε αυτό το στοιχείο να ληφθεί υπόψη. Θα είναι μια, ένα πολύ σωστό κανάλι να ακολουθήσουμε για να διαπιστώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Εάν όμως διαπιστώσουμε ότι οι φώκες δεν τρώνε το σολομό και ότι δεν φταίνε για τη μείωση του είδους και τρώνε μόνο ε, τα ψάρια τα οποία υπάρχουν σε εκβολές των ποταμών, τότε δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό και να ενισχύσουμε την ανασύσταση. Ε, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα διότι από, από αυτά τα στοιχεία εξαρτώνται και οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα εις βάθος όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουμε βάσιμες ε, πηγές πληροφόρησης, δεν έχουμε κατάλληλα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων και υπάρχουν και πολλά άλλα αμφιλεγόμενα στοιχεία ε, και όπως παραδείγματος χάρη η παράδοση της αρμοδιότητας για τα εσωτερικά ύδατα στην ε, Κομισιόν για να μπορεί να εποπτεύει και να ελέγχει αυτά, αυτούς τους, ε, αυτή την αλία. Θέλω λοιπόν να ακούσω και από εσά τι γνώμη έχετε για την παράδοση της αρμοδιότητος των ε, εσωτερικών υδάτων, ποταμίων υδάτων δηλαδή στην Κομισιόν. Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές αποφάσεις ε, για το μέλλον. E, και έχει και μεγάλη σημασία η καταγραφή αυτών των στοιχείων στα ημερολόγια πλοίων. Όταν έχουμε έναν αλιέα ο οποίος έχει ένα σκάφος 4-5 μέτρα, είναι πολύ μικρό και δεν, δεν κρατάει ημερολόγιο πλοίου Σε αυτή την περίπτωση μου φαίνεται ότι είναι παράλογη η επιβολή, ας πούμε, καταχώρησης, ε, διότι θα δημιουργήσει προσκόμματα στους, ε, στους συγκεκριμένους αυτούς μικρών σκαφών. Δεν είμαι εναντίον των μερολογίων ε, πλοίων, χρειαζόμαστε, τα χρειαζόμαστε για τους ελέγχους, αλλά υπάρχει και η αλία αναψυχής, η οποία δεν ελέγχεται και δεν υποπτεύεται καθόλου και δεν έχουμε ιδέα το τι γίνεται σε αυτό το τομέα ούτε έχουμε ιδέα εάν η αλία αναψυχή έχει επίπτωση γενικά στα αποθέματα του Σολομού. Όλα αυτά τα στοιχεία θέλω να τα αναφέρω στην ε, γνωμοδότησή μου και γι' αυτό ακριβώς θέλω να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριος ε, Χάντον. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ντοσχέ αυτό για τον εισηγητή, διότι η κατάσταση είναι λίγο ανησυχητική στη Βαλτική για το Σολομό. Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει υπογραμμίσει τους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής ικανοποιητικά. Όταν λέει ότι τα αποθέματα του Σολομού στη Βαλτική πρέπει να, να εκμεταλλευτούμε με βιώσιμο τρόπο εξασφαλίζοντας ε, την, βιο, την ποικιλία, την βιοπικιλότητα του Σολομού της Βαλτικής. Τα λέει πολύ σωστά. Αυτό που έχω εγώ να κάνω είναι δύο σύντομα σχόλια. Καταρχάς η παράνομη αλληλεία στη Βαλτική Έχω υποβάλει μια γραπτή ερώτηση, ένα γραπτό ερώτημα στην Κομισιόν επ' αυτού και είχα μια πολύ ικανοποιητική απάντηση από την Κομισιόν. Μου απάντησε η Κομισιόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε είναι γεγονός ότι γίνεται ε, σοβαρή παράνομη αλία, ένα σοβαρό ποσοστό παράνομης αλίας και αυτό έχει άμεση επίπτωση στα αλλιεύματα που επιτρέπουμε, διότι ξεπερνιούνται τα επιτρεπόμενα όρια λόγω της παράνομης αλλίας. Και αυτό επηράζει αποφασιστικά την ε, πολύ αρνητική κατάσταση των αποθεμάτων Σολομού πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και αυτό το στοιχείο να το αναφέρουμε στην έκθεση. Η Κομισιόν μας έχει πει ότι θα το, το στοιχείο αυτό το λάβει υπόψη ε, στην στρατηγική της του επόμενου έτους. Όπως ανέφερε ο εισηγητής και εγώ θέλω να το θίξω αυτό, είναι ο πληθυσμό των φώκεων. Οι φώκες πραγματικά έχουν, ε, είναι πολυπληθείς στην περιοχή αυτή και Εάν δούμε το ιστορικό υπόβαθρο, παλιότερα το κυνήγι της φώκιας ήταν τόσο έντονο που είχε μειωθεί ο πληθυσμός. Τώρα όμως μειώθηκε το κυνήγι της φώκιας και έτσι ανασυστάθηκε ο πληθυσμός τους και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει την αλήθεια στη Βαλτική διότι όταν πιάνουν τα ψάρια στη Βαλτική βλέπουν ίχνη ε, τραυμάτων από δαγκώματα φώκιας σε πολλά ψάρια. Εγώ υποστηρίζω την ε, επέκταση της άδειας ε, αλίας της φώκιας, κυνηγιού της φώκιας, προσωπικά, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ε, ε, εμπίπτει μέσα στο πεδίο ισχύω της, ε, ισχύως της γνωμοδότησης, διότι το βασικό δεν είναι ούτε οι φώκες ούτε οι κορμοράνοι, αλλά το, η αλληλεία του Σολομού και το γεγονός ότι η πραγματική αλληλευσή ξέπερνα τα επιτρεπόμενα όρια τα επιτρεπόμενα τάκ. Ε, γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του Σολομού για το μέλλον και αν δεν αναλάβουμε δράση στη Βαλτική ε, πολύ σύντομα δεν θα επιτύχουμε στο στόχο μας αυτό της διατήρησης και βιωσιμότητας του Σολομού. Ο κύριος Πούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συμφωνώ με τον προλαλήσαντα και τον εισηγητή με αυτά που είπα. Ότι χρειαζόμαστε σαφώς μία, μία αξιόπιστη ανάλυση της κατάστασης του Σολομού. ακούμε, μαθαίνουμε μόνο την, τα στοιχεία από την ΆΙΣΕΣ για την βιομάζα, ε, για και, και άλλες πληροφορίες που δεν εγγυώνται την επιβίωση και τη διατήρηση των αποθεμάτων. Πρέπει το πολιετές αυτό πρόγραμμα να βασίζεται στην βιώσιμη αλληλεία του <coughs> Σολομού, να εγγυάται τη βιώσιμη αλληλεία. Επίσης, δεν νομίζω ότι όλες οι παράμετροι επιπτώσεων και πάνω στην αλία του Σολομού έχουν αναλυθεί σωστά. Ε, παραδείγματο χάρη, οι συνθήκε, τα, τα, τα, τα ποσοστά των ε, ηχθειοτροφίων, η ηχθειοκαλλιέργεια του Σολομού, παραδείγματο χάρη. Ε, επίσης, ε, η το κυνήγι του σολομού από, από άλλα είδη ε, ή από πουλιά, από τους κορμοράνους παραδείγματο χάρη και από τα άλλα θηλαστικά τα οποία υπάρχουν στη Βόρειο Θάλασσα και στη Βαλτική. Ε, όλα αυτά δεν έχουν ε, αναλυθεί ικανοποιητικά και σωστά. ο πλησισμός των φώκιων, των θαλασσίων λεόντων και των κορμοράνων δεν είναι γνωστή, δεν έχουμε κάνει ποτέ καμία τέτοια ανάλυση και τι επίπτωση έχει το κυνήγι του Σολομού από τα άλλα είδη ε, θηλαστικών και πουλιών στην Βαλτική. Αλλά ότι υπάρχει επίπτωση υπάρχει. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι μια καταγραφή του αποθέματος πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε και τα, τους ε, νέους σολομούς, τα μικρά ψάρια, τα μικρά σε ηλικία ψάρια και ε, τα εσωτερικά ύδατα. Ε, και βεβαίως ε, ανάλυση στοιχείων για την παράνομη αλία. Όποιος έχει μία άδεια αλίας και ένα τάκ μπορεί να αλλιεύσει, αλλά ότι υπάρχει παρανομή, υπάρχει είναι γεγονό. Επίση, την αλληλεία αναψυχή και αυτή πρέπει να την υπολογίσουμε διότι η αλία, τα από την αλληλεία αναψυχής πρέπει να συμπεριληφθούν στα ΤΑΚ. Τώρα οι στόχοι τη Κομισιόν για το πολιετέ ε, πρόγραμμα βασίζονται στην ε, βιώσιμη αλληλεία, ε, διατήρηση της βιοπικιλότητας όλα αυτά πολύ σωστά και εκεί όπου υπάρχει ακόμα, όπου υπάρχουν ακόμα εξιοτροφία στο θα πρέπει να μειωθούν ε, μέσα σε 7 χρόνια οι ποσότητες αυτές. Οπότε θέλω και εγώ να ρωτήσω πώς θέλετε να βιώσουμε και να αγγιθούμε τη βιωσιμότητα του Σολομού θα θέλετε να ανακατέψουμε τον ε, Σολομό θα εξιοτροφία με τον άγριο Σολομό. Να μειώσουμε τον έναν υπέρ του άλλου. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα. Για, τα για το νομοθετικό πλαίσιο τώρα έχουμε τα ΤΑΚ, τα τεχνικά μέτρα και Εάν αυτά τα μέτρα δεν γίνονται σεβαστά διεθνώς, τότε η Κομισιόν θα πρέπει να παρέμβει. Θα πρέπει να επιβάλλει ε, κυρώσεις ε, διοικητικής και αλλιευτικής φύσης, αλλιευτικά και διοικητικά μέτρα δηλαδή, Θα πρέπει τώρα τα σκάφη αναψυχής, άμα θέλουν ε, να, η αλία αναψυχής ε, και τα σκάφη αναψυχής, εάν θέλουν να ψαρεύουν σολομό, να έχουν ειδική άδεια. Αυτό το, το είπαμε. Και επίσης τα μικρά αλλιευτικά σκάφη θα πρέπει να, εμπε, εμπίπτουν απόλυτα ε, στον, στις διαδικασίες ελέγχου κάτω από 10 μέτρα πρέπει να έχουν μερολόγιο πλοίου πρέπει να δούμε τώρα ποιο ποσοστό αναλογεί στα μικρά αλλιευτικά σκάφη 10% συν πλήν πόσο. Ε, εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της αλίας αναψυχής διότι και άλλα είδη όπως ο γάδος, όπως πολύ καλά ξέρουμε, μειώθηκαν τα αποθέματα του τόσο δραματικά, δεδομένου ήταν ελεύθερη αλία σε όλους. Ε, γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός, αλλά και οι σεμιτές συνθήκες, δίκαιες συνθήκες για όλους στην αλία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα της Κομισιόν για τη Βαλτική Θάλασσα είναι πολύ θετικό. Έχει πάρα πολλά ε, καλά στοιχεία τα οποία προσμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Παραδείγματο χάρη αναφέρεται στο Σολομό, σε όλο το κύκλο ζωής του Σολομού, αναφέρεται στην αλία αναψυχής, αναφέρεται την τεχνητή ανασύσταση και αντιστάθμιση του ελλείμματος του Σολομού στη Βαλτική, πολύ σωστό. Επίσης, η πέστροφα, αναφέρεται στη θαλάσσια πέστροφα. Έχουμε όμως και ερωτήματα και παρατηρήσεις για τους μικρούς Σολομούς και τους στόχους για τα μικρά ποτάμια προτείνεται 70%. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει στο πρόγραμμα δράσης για τη Βαλτική ότι πρέπει να είναι 80% το δυναμικό το, του μικρού Σολομού, του νέου Σολομού. Ε, γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορά στα ποσοστά. Και κάτι άλλο, είπατε ότι το δυναμικό μικρού Σολομού είναι το σημείο εκκίνωσης. Όμως ε, δεν αναφέρεται την ε, επιστροφή ε, των Σολομών στα εδάφια αναπαραγωγής, του αναπαραγωγικού Σολομού. Στα σουηδικά ποτάμια είδαμε μια ανησυχητική συμπεριφορά των Σολομών που επιστρέφουν για ανάντι, δηλαδή για αναπαραγωγή. Βρίσκονται εκτός ισορροπίας, δεν μπορούν να προχωρήσουν σωστά στα ποτάμια. Μια περίεργη συμπεριφορά που φαίνεται ότι κάτι δεν είναι καλά στους οργανισμούς των ψαριών αυτών. Επίσης, υπάρχει μία έλλειψη ε, στα, στους σολομούς αυτούς ε, θιαμίνης και βιταμίνης D. Υπάρχουν ορισμένα αντισυχητικά στοιχεία λοιπόν όταν εξετάσαμε τον αριθμό αλλά και την φυσιολογική κατάσταση των των... του αναπαραγωγικού σολομού που επιστρέφει στα ποτάμια. Λοιπόν, η αλληλεία αναψυχής είναι ένα πάρα πολύ ε, μικρό ποσοστό. Σύμφωνα με την ISIS, περίπου 23% των συνολικών αλλιευμάτων οφείλονται στην αλληλεία αναψυχής. Ε, και από απόψε Σολομού δηλαδή, πάρα πολύ λίγη η ποσότητα Σολομού αλλιεύεται από την αλληλεία αναψυχής. Γενικά η αλία αναψυχής, ανψυχής σε εισαγωγικά δηλαδή, γίνεται όχι από μένους αλείς, αλλά με δίχτυα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ατομική αλία, αλλά μέτρα δίχτυα τα σκάφη αυτά ρίχνουν ε, έξω από την περιοχή των 300 μέτρων σε απόσταση πάνω από 300 μέτρα από την ακτή. Και αυτά τα λιεύματα ξεφεύγουν κάθε ελέγχου. Δεν αναφέρονται, δεν καταγράφονται. Είναι κάτι πολύ σοβαρό λοιπόν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει φώκια η οποία, ή φώκιας που θα έτρωγε θα κατασπάραζε, θα πούμε καλύτερα, τόση μεγάλη ποσότητα σολομού όσο αυτή που μας ξεφεύγει ελέγχου από την αλία αναψυχής. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι να ε, συμπεριλάβουμε όλο τον κύκλο ζωής του, των ψαριών και στη θάλασσα και στα ποτάμια. Ωραία είναι όλα αυτά τα προγράμματα διαχείρισης και τα μέτρα διαχείρισης, αλλά το άρθρο 6, παράγραφος 6 λέει, εάν τα κράτη-μέλη δεν φροντίσουν τα μέτρα να είναι συμβατά με τους στόχους που θέτονται για τη Βαλτική, τότε η Κομισιόν θα λάβει μέτρα, εξαιρετικά, μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Όμως, το ερώτημα μου είναι, δεν θέλετε να κάνετε μια αξιολόγηση των μέτρων των κρατών μελών εξ αρχής, αντί να περιμένετε χρόνια για να κάνετε την αξιολόγηση εκ των υστέρων. Θα σταματήσω εδώ. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ ο κύριος ε, Καπάτσεκ έκανε μια διεξοδικότατη παρουσίαση για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μόλις τώρα μας έλεγε η κυρία Λεβίν ε, ότι ε, δεν έχει ληφθεί υπόψη το μεγεθό και το είδος των δικτυών ε, ούτε και ε, λάβαμε υπόψη τους, ε, τις φώκες θηρευτές και την επιρροή που έχουν στο απόθεμα Σολομού. Στην Σκοτία στην Άμποτη βλέπω πάνω στις, στους αμολόφους ένα τεράστιο πληθυσμό ε, από φώκες ε, που καταβροχθίζουν τους γεννήτορες που προσπαθούν ανάδρομα να ξανανεύουν ε, το ποτάμι για να αναπαραχθούν. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, στη Σκοτία έχουμε σοβαρά προβλήματα με ε, τα ελάφια. Είχαμε και ειδική επιτροπή και ολόκληρο πρόγραμμα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και ε, ο πληθυσμός ε, είναι υπέρ όλων των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος για τα ελάφια, για τις μέλισσες αλλά για τις φώκες είναι τόσο προστατευμένο το είδος που ούτε καν αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη λέξη φώκια με στις εκθέσεις της. Δεν ζητώ σφαγή του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Νομίζω ότι εκλογικός πώς θα ήταν αυτοκτονία από πλευρά μου. Αλλά καιρός δεν είναι να λάβουμε υπόψη ε, το ότι είναι θηρευτές οι φώκες και επιτίθενται σε ευαίσθητα αποθέματα όπως ε, ο Σολομός της ε, Βαλτικής. Γιατί συνεχίζει η Επιτροπή να αγνοεί αυτή τη διάσταση, μπορείτε να το εξηγήσετε. Ο κύριος Λάιτερ. Χαίρομαι που ξανάρθα στην Επιτροπή, που γύρισα στην Επιτροπή και ήρθα εδώ γιατί είμαι συντάκτη ε, μια σχετική έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Ακόμη δεν έχει γίνει η συζήτηση, άρα δεν μπορώ να σα μεταφέρω και την επίσημη θέση τη Επιτροπή. Θυμάμαι ότι την περασμένη φορά που ε, ψάρεψα εγώ έναν άγριο σολομό ήταν πριν από 35 χρόνια. Τελευταία φορά τότε είδα εγώ εκεί στο εξοχικό μου στη Σουηδία τον ε, Άγριο Σολομό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αν ε, ε, τελικά γίνει πραγματικότητα το σχέδιο ανάκαμψης του αποθέματος, μπορεί και να ξαναδώ Σολομό. Πάντως είναι σωστά τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα αποθέματα είναι χείρις της ποιότητας και επίσης τα ποσοστά επιστροφής είναι εξαιρετικά χαμηλά. Ε, δεν μπορούμε να δώσουμε μια ικανοποιητική εξήγηση γι' αυτό, αλλά αμφιβάλλω ότι φταίνε οι φώκες ε, μέσα στην Βαλτική, ξέρετε, μένουν κοντά στην ακτή και αν εξαφανίζονται στα ανοιχτά και δεν επιστρέφουν, πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος. Εγώ ε, συζήτησα με έναν καθηγήτη θαλάσσιας βιολογίας και μου έδειξε περίπλοκα στοιχεία για την αλυσίδα. Ποιος τρώει ποιον δηλαδή. Ε, γιατί οι φώκες δεν τρώνε μόνο ε, η διατροφική αλυσίδα είναι εξαιρετικά περίπλοκη και αρχίζει με το πλανκτόν. Η, στη Βαλτική είναι πολύ είναι η κρίση. Επίσης τώρα συζητάμε για την απαγόρευση ε, των φωσφόρων για αυτά τα προϊόντα, τα απορριπαντικά ε, που χρησιμοποιούνται για τα πλυντήρια πιάτων και άλλα. Ε, αυτό είναι σημαντικό ε, μέσα στην διατροφική αλυσίδα. Γιατί θα, το σπράου της Αρδελόρεγκα θα αυξηθεί πάρα πολύ αν ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Θα επηρεαστεί δηλαδή το πλανκτόν και θα διαταραχθεί ε, όλη η αλυσίδα πάντως. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα από επιστημονικής πλευράς και δεν θα καταλόγιζα εγώ όλα τα κακά στις φώκες. Ε, ε, και αν τα αφήσουμε τα πράγματα ήσυχα και δεν παρεμβαίνουμε, μάλλον θα ρυθμιστούν από μόνα τους. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Γιατί δεν επιστρέφουν οι γεννήτωρες, Αυτό είναι σημαντικό. Το άλλο στοιχείο που έχει σημασία και καλό θα ήταν να βρει μια νέα λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό είναι αυτή η ε, καταναγκαστική εισαγωγή ηχθιδίων σολομού ε, για ε, να ε, ενισχύσουμε τη βιομάζα. Μάλιστα, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει και αναπαραγωγή, να επιστρέψουν αυτά τα ψάρια, αλλά επιστρέφουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Όταν επιλογίζουμε όμως ε, τον φόρο, το ΤΑΚ, συγγνώμη, σε μεγάλο βαθμό συνυπολογίζουμε τα άγρια ψάρια και σκοτώνουμε τα ψάρια που θα μας βοηθούσαν να, που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν. για την εραστεχνική ε, αλία. Ίσως είναι παράλογο να περιμένουμε ότι όλοι θα ε, ε, υποβάλουν όλα τα στοιχεία αλλά χρειαζόμαστε μια καλύτερη γνώση για τα αλλιεύματα, ε, κυρίω για τα προβλήματα των δικτυών. Μπορεί να είναι αμυγό ειδικό πρόβλημα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πάντω για τους εραστέχνες ε, μπορούμε να έχουμε προσωρινά ή περιφερειακά κριτήρια υποβολή αναφορών, όχι να του ζητάμε να μα κοινοποιήσουν όλα τα στοιχεία, αλλά σε κάποια μέρη, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να υποβάλουν πλήρε ε, αναφορές για να ξέρουμε ακριβώ αν τηρούν τη δική του ποσόστοση ε, για την αλίευση του συγκεκριμένου είδους. Ε, όταν έχω περισσότερε λεπτομέρειες, ε, μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα σας ενημερώσω και πάλι. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια προς την Νομική Υπηρεσία. Καταρχάς, για την αλληλεία αναψυχή. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γιατί σε περιπτώσεις όπως ο ερυθρός τόνος, η αλληλεία ψυχής προσμετράται και προσμετρέται βάσει της ποσόστοσης, εντός της ποσόστοσης των κρατών μελών και σε άλλες περιπτώσεις όπως αυτή δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η αλληλεία ψυχής. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Προφανώς υπάρχει κάποια λογική εξήγηση την οποία θα ήθελα να μου εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσον αφορά την ερώτηση προ την νομική υπηρεσία, διάβασα το σημείο που προετοιμάσατε και θα ήθελα να μου εξηγήσετε ε, πιο αναλυτικά το εξή. Εσείς αμφισβητείτε το άρθρο 27, δηλαδή την παρέκκληση των ε, ε, εξουσιών που εκχωρούνται στα κράτη-μέλη για τα σημεία 6 έως 11. Και εμένα σε σχέση και με την πρόταση για το βασικό κανονισμό που υπάρχει ανάλυ, ε, κάτι αντίστοιχο μου εξέπληξε αυτό. Ε, θα μπορούσαμε να το ε, αντιπαραθέσουμε με το βασικό κανονισμό γιατί θα δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον νομικό πρόσκομα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μου το εξηγήσετε γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι η μεταφορά στο βασικό κανονισμό για τα εθνικά ζητήματα, το κατά πόσον ε, τα εθνικά μέτρα δεν τηρούνται σε συγκεκριμένε προθεσμίε, υπάρχουν τρία χρόνια, τρει μήνε, μπορεί να γίνει ανάκληση τη εκχώρηση και από εκεί και πέρα να αναλάβει τα ενία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω λοιπόν, λοιπόν πρώτα το λόγο στην νομική υπηρεσία και μετά το λόγο στην Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αληθεύουν αυτά που λέτε. Υπάρχουν ε, πολλές ομοιότητες με τον νέο κανονισμό, τον νέο βασικό κανονισμό και αναλύουμε τώρα το βασικό κανονισμό ε, στα πλαίσια της αναθεώρησης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Θα εκδώσουμε γνωμοδότηση σύντομα. Και θα ε, δίνουμε κάποια απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα που συνδέονται με το Σολομό της Βαλτικής. Λάβαμε γνώση της πρότασης αυτής νωρίτερα και έτσι μπορέσαμε να καταλάβουμε τον τρόπο σκέψης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγκυδε προφανώς ε, στην εκπόνηση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών για το πολιετές πρόγραμμα αποκλειστικά και μόνο μέσα από αυτόν τον λεπτομερή κανονισμό σε σχέση με την πρόταση για το Σολομό της Βαλτικής και λαμβάνοντας ε, υπόψη τις ε, κατευθυντήριες γραμμές της γενικής αρχικής πρότασης της Επιτροπής μέσα σε αυτή μας τη γνωμοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, δηλαδή σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριες ε, γραμμές όταν θα εκπονήσουμε το νέο βασικό κανονισμό αντί Αντίθετα, σε ποιο βαθμό ε, δεν θα χρειαστεί να τις εφαρμόσουμε για κάποια συγκεκριμένα είδη. Ο κύριος Κούν νωρίτερα αναφέρθηκε σε ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω. Πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί η Επιτροπή να αντικαταστήσει τις ε, δικές της πράξεις ε, κατεξουσιοδότησης όταν δεν μεταφέρουν και εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη επαρκώς ένα νομοθέτημα της Ένωσης. Αυτό το θέμα των πράξεων κατεξουσιοδότης θα μας απασχολήσει όταν θα επεξεργαστούμε τη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική για τον νέο βασικό κανονισμό, αλλά αυτό ισχύει και για το Σόλωμο, γιατί γνωρίζουμε γι' αυτό το είδος, το σύνολο των μηχανισμών, αλλά θα σχετίζεται και με ε, αυτό το προπαρασκευαστικό σημείωμα που είχαμε ε, προετοιμάσει, που είχαμε εκθέσει διάφορα άλλα ε, ζητήματα. Πάντως μην ανησυχείτε. Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο θα έχουμε γνωμοδοτήσει εμείς για την μελλοντική αναθεώρηση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής και άρα θα έχετε τα απαιτούμενα μέσα στη διάθεσή σας για να αξιολογήσετε επαρκώς τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια που θα πρέπει να υιοθετήσουμε μέσα στο νέο βασικό κανονισμό και αντίστροφα είπαμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να, εξουσιο... να αναθέσει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στα κράτη-μέλη κάποιες αρμοδιότητες για να αντικαταστήσει πράξη κατά εξουσιοδότηση όταν υπάρχει παραβίαση από πλευρά των κρατών μελών των κανονισμών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μοντεσί τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Πολλές ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να σχολιάσω ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν. Πολλοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη μιας σαφούς ανάλυσης των αποθεμάτων. Πόσο, πόσα είναι τα αποθέματα, τι επιπτώσεις περιπτώσεις ε, έχει το κυνήγι της Φώκιας ε, στο Σολομό, του Κορμοράνων, την ε, μικρή, το μικρό ποσοστό επιστροφής των γεννητόρων κλπ. Το θέμα είναι ότι εμείς βασίζουμε τις αναλύσεις μας στα καλύτερα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας πιστεύω ότι δεν μπορούμε σε βάσος να αναλύσουμε όλα αυτά τα θέματα που τέθηκαν. Ε, αλλά ορισμένα από τα αποθέματα των ποταμί, του ποτάμιου Σολομού είναι εκτός ε, των ε, βιο της δυνατότητας ε, ανασύστασης και πραγματικά είναι σε πάρα πολύ κακό σημείο τα αποθέματα του Σολομού. Είναι λοιπόν ε, ε, αναγκαίο να λάβουμε τα, τα μέτρα που πρέπει το ταχύτερο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δραματική. Για να μπορέσουμε να αγγιθούμε την ανασύσταση του αποθέματος και τη γενετική ε, ποικιλότητα και ακαιρεότητα του είδους. Γι' αυτό συμφέρον μας είναι να επέμβουμε το ταχύτερο και να διαχειριστούμε την αλία με μία μακροπρόθεσμη στρατηγική, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Και το πρώτο πρέπει να κάνουμε να μειώσουμε τα επιτρεπόμενα λιεύματα, Να μειώσουμε τα τάκ. Αυτό βεβαίως δεν θα μας εμποδίσει να συνεχίσουμε τις αναλύσεις μας σε συνεργασία με τα επιστημονικά όργανα, τους επιστημονικούς φορείς όσον αφορά τα ζητήματα που θέσατε, ε, τους λόγους για τους οποίους ε, οι γεννήτωρες Σολομή ε, δεν επιστρέφουν στην ποσότητα που θα έπρεπε δηλαδή για να αναπαραχθούν κλπ. κλπ. Η ICC πιστεύω ότι μελετά το λόγο του υψηλού ποσοστού θνησιμότητος αυτών των γεννητόρων και ε, παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος, όμως εμείς ε, έχουμε μεγάλη πίεση να εφαρμόσουμε μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω της κακής κατάστασης. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι καλύπτουμε και τις θαλάσσιες ζώνες και τις ποτάμιες σε αυτήν την ε, πρόταση. Ο Σόλομος χρησιμοποιεί και τις δύο αυτές περιοχές. Περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στα ποτάμια. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιοριστούμε στη θάλασσα μόνο και να προτείνουμε μέτρα διατήρησης προστασίας ή ανασύστασης σε μόνο για τις θαλάσσιες περιοχές. Γι' αυτό στο νέο αυτό πρόγραμμα προτείνουμε μέτρα ε, και για τη θάλασσα όπως παραδοσιακά κάνουμε αλλά και για τα ποτάμια. Ίσως δεν είναι σαφές στο σημερινό βασικό κανονισμό ότι εμείς λόγω της συνθήκης της Λισαβόνα στο άρθρο 3.1 Δέλτα μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε και τα ποτάμια. Λέει λοιπόν το άρθρο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την ε, την προστασία όλων των βιολογικών, ε, των έμβιων οργανισμών στις υδάτινες περιοχές, θαλάσσιες και ποτάμιες και γι' αυτό ακριβώς μέσα του άρθρου αυτού έχουμε συμπεριλάβει πλέον και τα ποτάμια στο πλαίσιο του προγράμματός μας. Λοιπόν, ε, τα κράτη-μέλη έχουν συναρμοδιότητα βεβαίως στη διαχείριση των ποταμίων υδάτων και των εμβίων όντων σε αυτά. Είναι μια νέα ευθύνη και γι' αυτό εμπίπτει στην πολιτική περιφερειοποίησης. Έχουμε δύο ειδών ε, μέτρων διαχείρισης. Ε, στη θάλασσα και στα ποτάμια. Διαχειριστικά μέτρα λοιπόν και για τη θάλασσα και για τα ποτάμια. Έχουμε τώρα τις αρμοδιότητες να εφαρμόσουμε ε, τους, ε, τα, μέτρα εκείνα τα οποία θα, ε, με τα οποία θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Γι' αυτό η Κομισιόν θέλει να εδραιώσει ένα διαχειριστικό πρόγραμμα με σαφείς στόχους και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα ε, που θα επιτρέψουν σε αυτά να επιτύχουν τους στόχους. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίσουν τα ΤΑΚ, τα τεχνικά μέτρα προστασίας ε, του ποταμίσιου Σολομού, βάσει των στόχων που θέτουμε. Βέβαια, οι Κομισιόν είναι οι σεματοφύλακες ε, της θάλασσας, των θαλασσών και παραμένουμε θεματοφύλακες και για την όλη εφαρμογή του προγράμματος και την εφαρμογή του κανονισμού. Και επίσης ε, μπορούμε να παρέμβουμε, να... Ε, αν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πολιτική μέτρα τα οποία δεν είναι συμβατά με το πρόγραμμα. Εάν λοιπόν ένα κράτος μέλος δεν σέβεται τα ΤΑΚ ε, ή όλα ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο μπορούμε να παρέμβουμε βάσει της ρήτρα παρέμβασης. Ε, λέγεται stepping close, clause, ρήτρα παρέμβασης. Είναι σωστό λοιπόν ότι έχουμε κάνει τις προβλέψεις μας για το διχειριστικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι ότου ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες ε, εποπτείες και ελέγχου από πλευράς κρατών μελών. Εμείς θα προχωρήσουμε με το προβλεπόμενο διαχειριστικό μας πρόγραμμα. Και ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρμογή των ε, ΤΑΚ. Αυτό το θέμα θα επανέλθει πολλές φορές στις συζητήσεις σας στο πλαίσιο της ε, αναθεώρησης. Step in. Uh, adopt αλλά αυτές οι αρμοδιότητες είναι σαφώς καθορισμένες ε, στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν έχουν μια συγκεκριμένη ε, προθεσμία αναθεώρησης. και το Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφωνούν για την κατεξουσιοδότηση πράξη, και αν υπάρχουν αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, τότε μπορεί να γίνει η υιοθέτηση από πλευράς κομισιών. Όλα λοιπόν τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο ρόλος του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να είναι εξασφαλισμένος με αυτό το πλαίσιο. Αλλά πιστεύω ότι θα τεθούμε υποδοκιμασία όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος περιφερειοποίησης. Γιατί έχουμε διαχειριστικό πρόγραμμα για το Σολομό, διότι κάθε ποτάμι έχει διαφορετικά στοιχεία και μία διαφορετική κατάσταση. Γι' αυτό ε, είναι δύσκολο να καταγράψουμε όλα τα στοιχεία, τις λεπτομέρειες και τις, ε, τα τεχνικά μέτρα για κάθε ποτάμι ξεχωριστά. Έχουμε λοιπόν δο, εξουσιοδοτήσει τα κράτη-μέλη να δράσουν για τα ποτάμια έχοντας ε, υπόψη τους την ποικιλία των συνθήκων που υπάρχουν στα ποτάμια. Και αναφέρθηκε επί μακρόν η αλία αναψυχής και μας ρώτησε πολύ σωστά η Κομισιόν γιατί ασχολούμεθα με το σολομό στην αλία αναψυχής και όχι με άλλα είδη ψαριών. Βεβαίως τον ερυθρό τόνο ενεργούμε μέσα στα πλαίσια του ICAT. Οπότε αυτό το θέτουμε στην άκρη, πάει αυτό. Αλλά εδώ για το Σολομό έχουμε μία πολύ ιδιαίτερη κατάσταση όπου η αλία αναψυχή συνεχώς αυξάνεται. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε τα μάτια μας και να συμπεριφερθούμε σαν να μην έχει επίπτωση η αλία αναψυχή στο Σολομό. Φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικότατη επίπτωση. Αυτή τη στιγμή οι επιστημονικοί φορείς υπολογίζουν ότι 35% των συνολικών αλλιευμάτων του Σολομού γίνονται μέσω της αλλίας αναψυχής. Όμως, αυτό δεν είναι απόλυτα αξιόπιστο στοιχείο, διότι δεν έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα για να ε, εγγυηθούμε την αξιοπιστία αυτού του ποσοστού. Όμως, η επίπτωση, η επίδραση της, αναψυχή, της ε, αλίας αναψυχής είναι σημαντική, χωρίς καμία αμφιβολία. Στο μέλλον ελπίζω να έχουμε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που μας χρειάζονται για την βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την αλία αναψυχής. Αυτό που προτείνουμε τώρα είναι ότι οι πάροχοι θα πρέπει να καταχωρηθούν, θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο καταχώρησης των σκαφών αυτών και των παρόχων αυτών των υπηρεσιών. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο γιατί δεν θα πρέπει να γίνει μια τέτοια καταγραφή και ότι τα αλλιεύματα από την αλλία αναψυχής πρέπει να συνυπολογίζονται στα ΤΑΚ. δεν μπορεί να ξεφύγει η αλληλεία αυτή, η αλληλεία αναψυχής από το διαχειριστικό μας πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα τις, ε, ε, την εκβολή, την, την απελευθέρωση του Σολομού στη θάλασσα ή στα ποτάμια είναι γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την βιοπικιλία του Σολομού και μας λέει ότι η απελευθέρωση πληθυσμού Σολομού ε, έχει αρνητική επίπτωση στο γενετικό υλικό του Σολομού. Πρέπει λοιπόν να ε, εφαρμόσουμε μία σταδιακή μείωση. Tomorrow. And we will be forecast also in the new ε, financial... των απελευθερώσεων αυτών ε, για να αντιστασμίσουμε την διατήρηση του του βιο, της βιοπικιλότητας του γενετικού υλικού και πρέπει να προβλέψουμε μέτρα αντιστάθμισης για τη μείωση αυτή των απελευθερώσεων, των ποσοτήτων που απελευθερώνονται. Όσον αφορά την παράνομη αλία, εδώ ανησυχούμε ιδιαίτερα από την πρόσφατη έκθεση της ΣΑΙΣΑΣ ε, για την παράνομη αλία. Πραγματικά μεγάλες ποσότητες και σοβαρή, σοβαρό ποσοστό παράνομης αλίας έχει διαπιστωθεί. Και ε, έχουν αναλάβει, έχουν υποσχεθεί τα κράτη-μέλη να σταματήσουν αυτήν την δραστηριότητα, αυτήν την παράνομη δραστηριότητα. Με διαφορετικά μέτρα, με κατάλληλα μέτρα. Ήδη το πρόγραμμα αναφέρει ορισμένα επιπλέον μέτρα ε, τα οποία θα ληφθούν, θα εγκριθούν στο μέλλον, αλλά εντωμεταξύ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την αυστηρή εφαρμογή των υπαρχόντων μέτρων καταπολέμησης και εμείς ως Κομισιόν αλλά και ε, οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρά αυτά τα μέτρα που υπάρχουν. Και θα εφαρμόσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα κοινό πρόγραμμα ελέγχων που θα ξεκινήσει στα μέσα του επόμενου έτους. Πρέπει να σας διακόψω γιατί ήθελα να το λόγο κάποιοι ευρωβουλευτές ε, όπως ο κύριος Στίβενσεν που λέτε ότι δεν απαντήσατε στις ερωτήσεις του. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε διότι πρέπει να σταματήσει η συζήτηση εδώ. Έχουμε άλλες δύο εκθέσεις και πρέπει να φύγουν οι συγητές. Πρέπει να τους δώσω το λόγο δεν δίνω σε άλλους το λόγο. Ε, θα συνεχιστεί η συζήτηση του ή άλλως κύριε Σλίτερ. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή γιατί έχει κόσμο που περιμένει όλο το πρωί και ακόμα δεν μπορέσει να μιλήσει και κάποιος εκ των εισηγητών πρέπει να φύγει. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλέ οι ερωτήσει χωρί απάντηση, αλλά εγώ δεν μπορώ να παρατείνω άλλο τη συζήτηση σήμερα. Κλείνει λοιπόν το θέμα αυτό, θα συνεχίσει η συζήτηση. Επιμένω, υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα και ε, στις επόμενες συζητήσεις θα έχουμε τη δυνατότητα να τα απαντήσουμε. Ο κύριος Αλαβράκος έχει παραχωρήσει τη θέση του πολύ ευγενικά στον κύριο Χάγκλοντ για να παρεύει, διότι πρέπει να φύγει σε ταξίδι ο κύριος Χάγκλοντ. Περνάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 14 και δίνουμε το λόγο στον κύριο Χάγκλοντ. Ένα τέταρτο το πολύ για να μείνουν τα υπόλοιπα 15 λεπτά της συνεδρίας στον κύριο Σολαβράκο. Κύριε Χάγκλοντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον συνάδελφο. Ε, πρέπει να φύγω σε λίγα λεπτά για το Παλέρμο για μια μεγάλη διάσκεψη. Ευχαριστώ για την ευελιξία που δείχνει ο κύριος Αλαβράκος. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια σύντομη παρουσίαση για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Που ονομάζεται... έκθεση ονομάζεται σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κατά εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της ΚΑΛΠ. Ε, η δική μου έκθεση τιτλοφορείται «Πρόσβαση στα ύδατα», αλλά ε, ο τίτλος του εγγράφου Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατά πολύ ευρύτερος, είναι εξαιρετικό το έγγραφο. Ε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά και συγκεκριμένα η κυρία Ρόντους σε σχέση με τον βασικό τεχνικό κανονισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα πορίσματα της εκθέσης και κυρίως της έκθεσης συγγνώμη, και τις ατέλειες ε, της ε, κοινή αλλιευτικής ε, πολιτικής Εντοπίζονται τα προβλήματα σε αυτό το επαναλαμβάνω εξαιρετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερόμαστε στα πολυετή σχέδια και λέμε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικά γιατί κατοχυρώνεται η μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποθεμάτων σε σχέση με τα ΤΑΚ. Η μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής το 2002 δεν κατάφερε να καταπολεμήσει την υπεραλίευση στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό το αναφέρει πολλές φορές το έγγραφό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη ε, το σύνολο των επιστημονικών στοιχείων για πολλά είδη, όπως και για το Σολομό, το είπαμε νωρίτερα. Αναφέρει ότι είναι σημαντικό να έχουμε και την οικοσυστημική προσέγγιση και οι Αμερικανοί και άλλοι Καναδοί και τα λοιπά έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με εμάς. Ε, Εν ώψη της επικείμενης αναθεώρησης ε, της ε, κοινή αλληλευτικής ε, πολιτικής είναι σημαντικό και ένα άλλο στοιχείο της έκθεσης, δηλαδή ότι εξακολουθούμε να έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την υπερδυναμικότητα του αλληλευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις μεταβιβάσιμες ατομικές ποσοστώσεις, αμφιλεγόμενο, πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα για πολλούς και άρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν χρειάζεται να εγκριθούν και άλλα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την υπερβολή υπερβολική ε, χωρητικότητα του στόλου ε, και επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα απόσυρσης ε, των αλληλευτικών σκαφών δεν έχει δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τώρα περνάμε στο, στη ζώνη των 12 μιλίων όπως ονομάζεται περιγράφεται μέσα στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρότι μάλλον είναι σύντομη αυτή η παρουσίαση Τα κράτη-μέλη και πολλοί εμπλεκόμενοι φορεί ε, ικανοποιούνται με τι τωρινέ ρυθμίσει. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αιτιολογηθεί μια αλλαγή. Τέλο πάντων, εν γέννη είναι πολύ χρήσιμο αυτό το έγγραφο, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή, ίσω όχι σήμερα, διότι δεν έχουμε και πολλούς βουλευτές εδώ. Ε, θα ήθελα τέλο να θέσω κάποια ερωτήματα υπόψη των συναδέλφων. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε με όλα αυτά τα χρήσιμα πορίσματα του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για να συντάξουμε μια καλή έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο και για να τροφοδοτήσουμε μέσα από αυτή την έκθεση τον προβληματισμό για την αναθεώρηση του βασικού κανονισμού. Χρονικός πώς ε, ε, τον Ιανουάριο θα είμαι σε θέση να καταθέσω κάποιο είδους έγγραφο εργασίας. Θα επιταχύνουμε τη διαδικασία για να κινηθούμε ταχύτερα από τι ε, ε, διαπραγματεύσει για τον τεχνικό βασικό κανονισμό, με στόχο βεβαίω να συμπεριληφθούν ε, στη νέα αναθεωρημένη εκδοχή του βασικού κανονισμού και θέση του Κοινοβουλίου, δηλαδή να καλυφθούν οι στόχοι που θελήσαμε εμεί να εισαγάγουμε σε αυτό το έγγραφο, όπω και στην έκθεση για την πράσινη βίβλο που συνέταξε η κυρία Πατράου Νέβε θα πρέπει να ε, υπολογιστούν τα στοιχεία, οι προτάσει που κάνουμε για την δημοσιονομική πλευρά της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Νομίζω ότι μπορώ να κλείσω εδώ την παρουσίασή μου και με ενδιαφέρει να ακούσω ε, το πώς τοποθετούνται οι συνάδελφοι σε σχέση με τα τόσο ενδιαφέροντα στοιχεία της έκθεσης και ε, ε, ανυπομονώ για την συνέχεια της ε, ενδιαφέρουσας αυτής της συζήτησης. να δούμε τους ε, συναδέλφους αν θέλουν το λόγο. Βέβαια είναι πολύ λίγοι. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Χάτλουν, το θέμα αυτό συνδέεται με τον ε, βασικό κανονισμό ε, και θα πρέπει να προηγείται η έκθεσή σας της έκθεσης της κυρίας Ρόντουστ. Βεβαίως είναι απαραίτητο και πρέπει να υπάρχει και μια λογική στις εργασίες ε, της Επιτροπής. Κύριε Πένας, ούτε και εγώ θέλω να μακρηγορήσω γιατί ξέρω ότι βιάζεστε και ο κύριος Αλαβράκος πρέπει να μιλήσει στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Πένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Όπως γνωρίζετε η έκθεση αυτή ε, θέλει να συμπληρώσει ούτως ή άλλως ε, δημοσιεύσεις ε, που έχουμε στο βασικό κανονισμό και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 35 του βασικού κανονισμού που ζητά αξιολόγηση των πολιτικών διατήρησης και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των ελευτικών πόρων και αυτό το έχουμε και στο άρθρο 17 που ζητά έκθεση για την εφαρμογή του κανόνα και των 12 μιλίων. Νομίζω ότι ο εισηγητής πολύ σωστά συνόψισε τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αξιολόγηση που κάναμε και για τις δύο θεμελιώδεις πολιτικές, ε, τη διατήρηση και την εκμετάλλευση του στόλου, περιλαμβάνει κάποιες θετικές πτυχές, κάποιες βελτιώσεις. Ίσως η πιο σημαντική βελτίωση χωρίς αμφιβολία είναι η αξιολόγηση των πολιτικών σχεδίων που όλοι αναγνωρίζετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη ζωστή κατεύθυνση αλλά χωρίς να είμαστε απεσιόδοξοι και χωρίς να λέμε ότι τα πάντα ήταν καταστροφή, υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις και υπάρχουν δύο πτυχές όμως της ε, πολιτικής διατήρησης, στην οποία δεν επετεύχθη μεγάλη πρόοδος. Από το 2012 και μετά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Το γνωρίζουμε εδώ και νέα χρόνια και η νέα μας διαπίστωση είναι ότι η πρόοδος που επετεύχθη για το στόχο αυτό στα τελευταία 9 χρόνια ήταν πάρα πολύ αργή. Πρόκειται για μια προφανή διαπίστωση. Έγιναν μεν κάποια θετικά βήματα, αλλά πάρα πολύ αργά και πολύ ε, ε, καθυστερημένα. Επίσης, το άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν βελτιωθήκαμε ε, πολύ σημαντικά στις γνώσεις μας για τα αλλιεύματα. Έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ε, αλλιευτικών προσπαθειών και ειδών για τα οποία δεν γνωρίζουν οι επιστήμονες σχεδόν τίποτα. Είμαστε ορισμένες φορές βυθισμένοι στο σκοτάδι και προχωρούμε στα τυφλά διότι γίνονται πάρα πολύ λίγα και γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα και ε, ελάχιστα, ε, αν όχι και μηδενικά στοιχεία για πολλά από τα είδη. Η πρόοδος λοιπόν για τους μακροπρόθεσμους στόχους είναι πάρα πολύ αργή και εξακολουθούμε να δυνατούμε να έχουμε μία κατάλληλη επιστημονική βάση για να διαχειριστούμε με καταλληλότερο τρόπο τα είδη μας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση του στόλου, και πάλι ο εισηγητή πολύ σωστά ανέλησε την κατάσταση, διαθέτουμε μια πολιτική η οποία επιφανειακά φαίνεται ότι λειτουργεί, αλλά στην πράξη ούτε καν μπορούμε να αξιολογήσουμε αντικειμενικά κατά πόσον υπάρχουν ε, σωστά στοιχεία και υπάρχουν και αρκετές ενδείξεις ότι δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Να εξηγήσω τι εννοώ. Εάν δούμε την πρόοδο στην πολιτική διαχείριση των στόλων μέσω των παραμέτρων που την καθορίζουν, δηλαδή κινητήρια, μοχλός και ταχύτητα, τεχνικώς λειτουργεί η πολιτική. Γιατί σε αυτές τις παραμέτρους έχουμε μειώσει την ουσιαστική δυνατότητα, την ονομαστική δυνατότητα και όλα τα κράτη-μέλη είναι εντός των ορίων που καθορίζονται. Στη θεωρία λοιπόν όλα βαίνουν καλώς. Γνωρίζουμε όμως ότι Καταρχάς, αυτές οι παράμετροι βάσει των οποίων καθορίζεται η παρούσα πολιτική των στόλων δεν λαμβάνουν υπόψη την ε, τεχνική πρόοδο των σκαφών, επομένως είναι λανθασμένη η ένδειξη της πραγματικής ισχύω και της ε, δυνατότητας αλίευσης των σκαφών. Και δεύτερον, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα διότι στην πράξη δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αντικειμενικά εάν υπάρχει υπερβολική αλίευση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ έμεσε ενδείξει που καταδεικνύουν ότι υπάρχει υπεραλίευση. Παραδείγματο χάρη, ποσοστά δραστηριότητα ε, με αριθμό ημερών ε, ε, ετησίων πολύ χαμηλέ, δηλαδή υπάρχουν δυνατότητε που δεν χρησιμοποιούνται, ποσοστά θνησιμότητα ε, ειδών ε, που καταδεικνύουν ότι υπάρχει υπεραλίευση σε κάποια είδη, ε, χαμηλή λειτουργικότητα σε πολλοί στόλους που μπορεί μεταξύ άλλων να οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχει και υπεραλίευση. δεν είναι λοιπόν αποτελεσματική η θεωρία στην πράξη, είναι μόνο στη θεωρία αποτελεσματική. Όσον αφορά το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι παρέκκληση στην αρχή της ελεύθερης πρόσβασης και θα πρέπει να εξετάσουμε και να αιτιολογήσουμε κατά πόσον πρέπει να διατηρηθεί αυτή η παρέκκληση. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία λήφθησαν υπόψη. Καταρχάς, στη διαδικασία διαβούλευσης δεν ήταν με νομόφωνη απόφαση, αλλά υπήρχε μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών και ενδιαφερομένων, η οποία ήταν υπέρ της ε, συνέχισης αυτής της παρέκκλησης των 12 μιλίων. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο σημείο. Ε, επικρίνεται αυτή η πολιτική από όλε τις πλευρές και επιτέλους υπάρχει κάτι το οποίο δεν επιχρίνουν οι πάντες. Επομένως αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Και επίσης αυτά τα 12 ναυτικά μίλια ε, στην πραγματικότητα παρά το γεγονό ότι κάθε κράτος μέλο μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί, να το ε, τηρήσει για κάποια σκάφη, για κάποια όλα, αποτελεί ένα καλό εργαλείο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε κατά κάποιο τρόπο τους τοπικούς στόλου, ιδίω τους μικρότερους στόλου όχι άμεσα, αλλά έμεσα αυτός ο κανόνας των 12 ε, μιλίων είναι τμήμα της όλης θεωρίας της ευνοϊκής μεταχείρισης προς τους μικρότερους τόλους. Επομένως, θεωρούμε για αυτούς τους δύο λόγους ότι αυτή η συνέχιση της παρέκκλησης ε, στην αρχή της ελεύθερης πρόσβασης είναι αιτιολογημένη. Θέλετε το λόγο κύριε Χάγκλουντ. Όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένος και θα φύγω για το Παλέρμο. Να περάσετε καλά, λέει η πρόεδρος. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα, τελειώσαμε με το σημείο 14 και να περάσουμε στο σημείο 13, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σαλαβράκο που παραχώρησε τη θέση του στον κύριο Χάγκλουντ. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την ε, ε ανακοίνωσή σας για τη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτική. πολιτικής. Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο διότι η σύγκριση του κύριου Χάγκλουντ είναι κοινή και πολλά από εισαγωγικά στοιχεία ταιριάζουν και στην έκθεση τη δική μου και επομένω δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Άλλωστε είμαστε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων και έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Ε, ενδιαφέρον κυρίως για την εξέλιξη της εκθέσεως είναι το γεγονός ότι η νομική υπηρεσία όπως μας είπε συντόμως θα έχει γνωμοδοτήσει πάνω στο νομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε ιδιαίτερα στο θέμα των 12 μιλίων και στο θέμα της αρχής της επικουρικότητας καθόν τρόπων θα ισχύσει στα θέματα των αλλιευμάτων διότι είναι προφανές ότι στην αλληλεία προχωρούμε πολύ περισσότερο σε μια πολιτική ένωση από ότι στην όλη Ευρώπη γενικότερα. Ε, είναι η τρίτη φορά βεβαίως ιστορικά στα 30 χρόνια της ιστορίας της ε, κίνησης αλληλευτικής πολιτικής που επανεξετάζεται το θέμα αλλά στην ουσία θα πρέπει να πούμε πράγματα που διαπιστώσαμε και πράγματα που, ε, για τα οποία έχουμε ερωτηματικά. Η, πρώτη διαπίστωση την οποία έχουμε είναι ότι χαιρόμεθα ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ε, σε συζητήσεις που κάναμε με αλληλείς είδαμε ότι ε, είναι εναντίον της παράνομης ε, αλλιέ και εναντίον του τρόπου αλλιεύσεως μετράτες ιδιαίτερα το βράδυ που πολλές φορές βάζουν ένα τενεκέ από ό,τι μου είπαν στην κεραία τους ώστε να μην ενιχνεύεται από το σύστημα παρακολούθησης τύπου Βίγκο και οργώνουν τη θάλασσα και την καταστρέφουν, καταστρέφουν τον βυθό. Είδα με συζητήσεις που έκανα τόσο με συνδικαλιστικά όργανα όσο και με μονομένους ότι η γενική τάση είναι αποδοκιμασία σε αυτή τη καταστάση. Τα ερωτηματικά τα οποία θέτω έτσι σύντομα είναι ότι στην ανακοίνωση γίνεται λόγος ειδικά για τη διαχείριση των οικείων στόλων της παράκτειας και μικρής Ε, θα ήθελα να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση γιατί σύμφωνα με τα όσα είδα η μεταβίβαση των ποσοστώσεων δείχνει μια φανερή πρόθεση βέβαια να ανοίξουμε την αγαρά αλλά για πολλούς με τους οποίους ομίλησε θεωρούν ότι πλήττονται οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή αιλία ενισχύεται ο συγκεντρωτισμός και θα έχουμε ψαράδες που θα έρχονται να ψαρεύουν ε, εις βάρος των παράκτιων αλλιέων. Αυτό ίσως δεν βοηθάει και στην ε, βιωσιμότητα των πόρων. Ένα δεύτερο ερωτηματικό το οποίο μου έθεσαν ε, είναι πώς θα επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ αλλιέας μικρής και μεγάλης κλίμακος ώστε να επιτρέπεται σε όλους να αλλιεύουν. Μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ανάλογα με την περιοχή ίσως πρέπει να υπάρχει και να έχει μια ε, και πρακτική αλλά και επιστημονική προσέγγιση ε, στην πρακτική των απορρίψεων. Στην πρακτική των απορρίψεων εκείνο το οποίο από την άλλη πλευρά διεπίστωσα είναι ότι υπάρχει και δυσκολία να ελέγχονται αλλιείς που δεν πετάνε τα ψάρια πίσω στη θάλασσα από την άλλη πλευρά υπάρχει για τους ίδιους τους αλλιείς ένα πρόβλημα επιπλέον αποθηκευτικού χώρου που θα χρειαστεί μέσα στο σκάφος και αυτό οπωσδήποτε στην πράξη θα έχει ένα πρόβλημα ανοιχνεύσεώς τους και παρακολουθήσει τους από πλευράς ας το πούμε εντός εισαγωγικών αστυνομεύσεως. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η μελέτη της ψυχολογίας του κλάδου για τη τελική ανάλυση από αυτό εξαρτάται η αποτελεσματικότητα ενός μέτρου. Ε, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για συνοδευτικά μέτρα που θα ακολουθήσουν το μέτρο αυτό και θα ήθελα να εξειδικεύσουμε ποια είναι αυτά τα ε, μέτρα. Ε, πιο κάτω θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, ιδίως στη Μεσόγειο, εκτός από την έλλειψη στοιχείων είναι συχνό φαινόμενο η επικάλυψη των αποθεμάτων λόγω της μεγάλης έκθεσης των διεθνών υδάτων και αυτό επηρεάζει σοβαρά την εφαρμογή του μοντέλου αυτού. Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή γι' αυτό παρακαλώ σημειώστε το για να έχουμε την ε, γνώση και την εμπειρία σας πάνω στο θέμα. Ιδιαίτερα χαιρετίζω βεβαίω την πρόταση τη Επιτροπή για την θέσπιση πολιετών σχεδίων διαχείριση ω μέσο αντιμετώπιση τη παραλίευση. Ωστόσο, θεωρώ ότι κάποια σημεία παραμένουν εκκρεμή και είναι απαραίτητη μια περαιτέρω εμβάθυνση για να θέσουμε πιο συγκεκριμένα μέτρα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα σε σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Θεωρώ ότι οι αλληλείς θα πρέπει να έχουν ένα κεντρικό ρόλο στη συνδιαχείριση και στο σχεδιασμό αυτών των σχεδίων διαχείρισης ε, και ως εκ τούτου θα πρέπει ίσως να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένους τρόπους για να ενισχυθεί η συμμετοχή των εκπροσώπων των αλλιέων στο θέμα. Ε, επίσης ε, θα ήθελα να δούμε την περιφερειοποίηση να την εξειδικεύσουμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα επιτευχθεί, με ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα συμπεριληφθούν οι αλλιείς στη διαδικασία διατήρηση τη βιωσιμότητα των αλλιευμάτων και να προσέξουμε και την κοινωνική διάσταση του θέματος διότι το επάγγελμα της αλληλείας γίνεται όλο και λιγότερο ελκυστικό για τους νέους έχουμε μια αφέμαξη νέων αλλιέων και ίσως θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα στους αλληλείς ε, που θα αποτελέσει κίνητρο παραμονής του στη θάλασσα. Ε, για τις ηχθιοκαλλιέργειες ε, το θέμα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, ίσως είναι και πιο επιστημονικά ε, αντιμετωπίσιμο και από πλευράς ε, ε των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Ε, για να μην ε, φάω περισσότερο χρόνο σταματώ εδώ και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία για να δώσουμε μια καλή έκθεση κατά το δυνατόν. Ευχαριστώ. Ε, Thank you. Ε, Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Σαλαβράκο. Είναι δύσκολο βέβαια να συζητήσουμε αυτήν την ανακοίνωση επειδή καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε ένα σημείο μόνο και δι στην πρόταση του TFC για τις ε, αλλιευτικές παραχωρήσεις, τις μεταβιβάσιμες ατομικές ποσοστώσεις. Αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι θα βοηθήσει και τους παράκτιους τόλους, τις παράκτιες κοινότητες και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να υποστηρίξουν τους μικρούς ε, αλληλείς, ε, την, ε, τις και γενικά την αλληλεία μικρής κλίμακος μέσω του, ταμείου, του Κοινοτικού Ταμείου Αλίας. Είναι πολύ σωστό λοιπόν να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά τα οικονομικά κίνητρα, τις μεταβιβάσιμε ατομικές ποσοστώσεις. Ε, πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες μας ε, θέλουν να ε, μην διακυβεύεται η ισορροπία των ε, ειδών, των ψαριών, έτσι ώστε μία αλληλεία η οποία είναι βιώσιμη και ικανοποιητική θα πρέπει να ενισχύεται έναντι μια άλλη η οποία είναι αρνητική, καταστροφική. Θα πρέπει όμως να εφαρμόσουμε και μέτρα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε αυτή τις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα επωφεληθούν από αυτές τις ποσοστώσεις, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν την πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό το στοιχείο λείπει από την πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή η διαχείριση της κατανομής των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων. Αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσον της κατανομής, έτσι ώστε όλη η αλληλεία που θα έχουμε να είναι αλληλεία ήπιων επιπτώσεων, να μην είναι αλληλεία η οποία να είναι περιβαλλοντικά ε, βλάψιμη, επιβλαβής, συγγνώμη, επιβλαβής. Πρέπει λοιπόν να ε, αναφέρουμε τις αρχές ε, της βέλτιστης πρακτικής. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι σε άλλους τομείς όπως τις εξορίξεις παραδείγματος χάρη εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Όμως εδώ περισσότερο η πολιτική μας βασίζεται στις ε, παραδοσιακές ε, ε, πολιτικές αλίες, στα παραδοσιακά αλιεύματα. Αυτές λοιπόν οι ποσοστώσεις, μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις έχουν ως στόχο να κάνουν μια ορθολογική διαχείριση της κοινοτικής αλίας έτσι ώστε να είναι ήπιον επιπτώσεων. Η Κομισιόν, κύριος Πένας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω και του δύο μιλητέ πολύ θετικέ οι παρεμβάσει του. Αυτό που έχει σημασία κυρία Πρόεδρε είναι να υπενθυμίσουμε λίγο ποιο είναι ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την ανακοίνωση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα σημαντική η συζήτηση αυτή τη ανακοίνωση. Διότι παρά το γεγονό ότι δεν είναι νομική φύσεω, έχει πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι ε, υψίστης σημασία, ε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι νομοθετικής φύσεως, για όλη την μεταρρύθμιση. Γι' αυτό ακριβώς και κάναμε αυτή την ανακοίνωση. Την ανακοίνωση, αν μου επιτρέψετε να σας το εξηγήσω, την κάναμε για τρεις λόγους. Καταρχάς, διότι πολλά από τα σημαντικά στοιχεία για το συνεκτικό πακέτο μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής δεν είναι θέματα νομικής φύσεως. Δεν θα τα βρούμε στο βασικό κανονισμό, ούτε στον κανονισμό για τη διαχείριση των αγορών, ούτε στον κανονισμό του Διαρθρωτικού Ταμείου. Ωστόσο, πρέπει να τα συζητήσουμε και βεβαίως παρά το γεγονός ότι δεν είναι νομικής ε, φύσεως είναι σημαντικά και παρά το γεγονός ότι δεν είναι νομικής φύσεως εδώ, τώρα, σε αυτή τη νομική βάση μπορεί να γίνει νομικής φύσεως σε άλλες νομικές βάσεις στο μέλλον να εξηγήσω δύο από τα θέματα τα οποία ανέφερε ο εισηγητή και μου φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικά. Καταρχά, το θέμα τη βελτίωση των δεδομένων και των επιστημονικών στοιχείων και δεύτερον, το θέμα τη κοινωνική διάσκαση ε, για τα αλληλευτικά σκάφη. Δύο θέματα τα οποία δεν έχουμε στι νομοθετικέ προτάσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα θέλαμε να συζητηθούν και στο περιθώριο τη απόφαση των νομικών θεμάτων θα θέλαμε οι συνομοθέτε να εκφράσουν και την άποψή του επ' αυτών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά στην ανακοίνωση. Δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η ανακοίνωση είναι το γεγονός ότι τα νομικά κείμενα τα γνωρίζουμε, ξέρουμε και με, από το παράδειγμα της περιφερειοποίησης ότι δεν είναι ε, αυτοεξηγούμενα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στα κείμενα, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με νομική ορολογία και πρέπει να επεκταθούμε για να δώσουμε την εξήγηση. Η ανακοίνωση επίσης θέλει να καθορίσει ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο ε, στο οποίο τα διάφορα τμήματα του πάζουλ αυτής της ε, μεταρρύθμισης θα μπορέσουν να συνενωθούν και να υπάρχει ένα κοινό θέμα. Ε, δεν είναι μόνο δυνατόν να πάρουμε την πρόταση για τις αγορές για να ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση οδεύουμε. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα μεμονωμένα. Εξηγούνται όλα πολύ καλύτερα σε ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εξηγούμε ποιες είναι οι βασικές κατευθυντήρες γραμμές για το θέμα αυτό. Αυτό ήταν ο στόχος μας με την ανακοίνωση. Τώρα επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε να επικεντρωθώ λίγο καλύτερα στα δύο θέματα στα οποία αναφέρθηκε και ο εισηγητή και ενδιαφέρουν νομίζω όλου μα. Η βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων. Εδώ υπάρχουν κάποια νομικά στοιχεία, κάποια οικονομικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν είναι νομική φύση και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί παραδείγματα, ετοιμάζει ένα σχέδιο για τη μελτίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που αποτελείται από αρκετά στοιχεία. Ένα ουσιαστικό στοιχείο είναι ε, η στάση μας προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να συλλέγουν τα βασικά δεδομένα για την ε, υποστήριξη των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Αυτό δεν το έχετε δει ακόμα, αλλά ε, θα το δούμε στον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Στο δημοσιονομικό κανονισμό υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την χρηματοοικονομική στήριξη στα κράτη-μέλη για τη συλλογή δεδομένων, των βασικών δεδομένων. Επιπλέον, στον κανονισμό αυτό θα δείτε ότι θα υπάρχει και μια γραμμή υποστήριξη ε, για τα σχέδια συνεργασίας μεταξύ του κλάδου και των επιστημόνων. Αυτό θα τύχει οικονομικής ενίσχυσης και υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε οικονομικά ούτε νομικά. Υπάρχει για παράδειγμα το πώς ε, θα οργανώσουμε τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτουμε σε επιστημονικό επίπεδο στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι περιορισμένοι, προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του συστήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον ICE, το CTFS, που σε μεγάλο βαθμό έχουν αλληλεπικάλυψη ε, εργασιών. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί ο συντονισμός του συστήματος, να βελτιωθεί η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο, ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τους ελάχιστους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας από επιστημονική σκοπιά. Και επίσης θέλουμε να έχουμε και μια πολιτική η οποία δεν θα είναι νομική, θα ε, βοηθά ώστε οι ευρωπαϊκοί ερευνητικοί οργανισμοί να μπορούν να διαθέτουν περισσότερους ανθρώπινους πόρους, να προσλαμβάνουν νέους επιστήμονες και να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη βάση που έχουμε σε ανθρώπινο δυναμικό για την εκπόνηση αυτών των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο το οποίο έχει μεν κάποιες νομικές πτυχές, αλλά πηγαίνει και πολύ περαιτέρω και αυτό ακριβώ αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε. Ήγηκε η ώρα λοιπόν εδώ το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο να συζητήσει τα θέματα αυτά. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της κοινωνική διάσταση. Μας λέγεται και προφανέω ότι το θέμα της κοινωνικής διάστασης δεν είναι προφανές ε, στις ε, προτάσεις. Υπάρχουν πολλά στοιχεία όμως της κοινωνικής διάστασης που ε, δεν επιτρέπουν για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει γιατί άπτονται μια άλλη νομική βάση, όχι τη νομική βάση που έχουμε εμεί εδώ. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που δεν θα δούμε εμεί εδώ στην κοινωνική διάσταση, αλλά αποτελούν τμήμα του σχεδίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τμήμα τη ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση, για παράδειγμα, έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τη κύρωση ε, τη σύμβαση ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασία για τις συνθήκες εργασία στα λιευτικά σκάφη. Πρόκειται για μια σύμβαση ε, του 2007 που ακόμα δεν έχουν κυρώσει όλα τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το αναφέρουμε αυτό, να δούμε πότε θα κυρωθεί αυτή η σύμβαση από όλα τα κράτη-μέλη, πότε θα τεθεί πλήρω ισχύ και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συζητήσουμε και τι συνέχεια θα δοθεί στο θέμα αυτό, ώστε να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις της σύμβασης σε κοινοτικό δίκαιο χωρίς να γίνει απαραίτητα στην νομική βάση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Πρώτη και ε, παρόλα αυτά για ένα σημαντικό πυλώνα της αλληλευτικής πολιτικής που πρέπει να συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτό. Για την ερώτηση της κυρίας Λεβίν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε γιατί δεν ε, περιλαμβάνεται αυτό το στοιχείο και δεν έχει δίκιο κυρία Λεβίν, δεν αναφέρουμε τίποτα γι' αυτό. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όπλο της κατανομής της μεταβίβασης των ατομικών ποσοστώσεων ως ένα εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέψει να ευνοούσουμε τις πιο βιώσιμες ε, αλλιευτικές ε, ε, δυνατότητες ή ε, αυτές οι οποίες είναι πιο ενδιαφέρουσες από κοινωνική σκοπιά. Ο λόγος για τον οποίο δεν προτείναμε τίποτα είναι γιατί γίνεται ένας παραδοσιακός καταμερισμός εξουσιών, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, υπό την εξή έννοια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει το σύστημα κατανομής τάκ και ποσοστώσεων μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα όμως, το τι κάνει κάθε κράτος μέλος με τους πόρους του αυτό παραδοσιακώ είναι αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να σεβαστεί αυτό τον καταμερισμό των εξουσιών και μάλιστα σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε εδώ στο Κοινοβούλιο, πολλοί από εσά είπαν γιατί να μην συμπεριλάβουμε και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα κράτη-μέλη κάποια υποχρέωση ώστε να αφιερώνεται ένα σημαντικό τμήμα των ε, ποσοστώσεών τους σε αλληλευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι πιο βιώσιμες. Δεν έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν εσεί ω συνομοθέτε το προτείνετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Δεν το προτείναμε όμω, διότι θεωρούμε ότι αυτό παραδοσιακά άπτεται των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σα πω ότι εν γέννη στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη. Ε, διστάζουν πάρα πολύ και θέλουν να υπάρχει αυτή η εξουσία σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα χαράς να τα συζητήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλαβράκο, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πέρασε και η ώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την παρουσία σας εδώ και σας παρακαλώ στις 3 ακριβώς να είστε στην ώρα σας γιατί έχουμε ακρόαση και θα ήθελα τουλάχιστον να έχουμε κάποιους ε, στην αίθουσα διότι Αλλιώς θα είναι άσχημο το θέμα που θα έχουμε εδώ στην αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Πέρασε η συνεδρίαση. Τα λέμε στις 3.